Uh, Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους εκπροσώπους ανωτέρου επίπεδου της Ιταλικής Προεδρίας. Πρώτα απ' όλα την κυρία Φεντερίκα Γκουίντι, που είναι Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, και τον κύριο Αντωνέλο Τζακομέλη, που είναι Υφυπουργός για τις τηλεπικοινωνίες στην Ιταλία. Ένα θέμα με το οποίο ειδικά ασχολείται ο κ. Τζακομέλη. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τους επισκέπτες μας. Η κυρία Φεντερίκα Γκουίδη, η Υπουργός, Αποφύτησε στην νομική από το Πανεπιστήμιο και από την αρχή της εμπορικής της, της ε, της εμπειρίας ασχολήθηκε με την βιομηχανία, με τους νέους επιχειρηματίες επίσης για τέσσερα χρόνια. Ήταν και πρόεδρος της κάτι Ενέργεια στην ε, Βολονία είχε επίσης, ε, στην Πολωνική, είχε επίσης και άλλες ε, σημαντικές θέσεις. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας, εσάς που θα εκπροσωπείτε την τελική Προεδρία τους επόμενους μήνες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα η βιομηχανοποίηση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βιομηχανική πολιτική, και πιστεύουμε ότι αποτελεί και μία συνέχεια με τον επίτροπο που είχαμε μέχρι πριν από λίγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδιο για αυτά τα θέματα, οπότε και αυτός Ιταλός και τώρα είναι εδώ μαζί μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι καλύτερα να μιλήσω τώρα Ιταλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Μπούζεκ ε, και αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που ε, συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ κυρίως για το γεγονός ότι μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τα θέματα του Υπουργείου μου. Και θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα της ενέργειας, της ανταγωνιστικότητας που ε, βεβαίως και έχουν σχέση με, τις, ε, με την ψηφιακή τηλεπιδιονία επί το οποίο όμως θα τοποθετηθεί ο κύριος Τσακομέλη ο Υφυπουργό. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω κάποιες σύντομες αρχικές παρατηρήσεις. Καταρχήν θέλω να πω ότι ε, προσπαθήσαμε να εστιάσουμε τις ε, δραστηριότητές μας ε, σε συγκεκριμένα προγράμματα φιλόδοξα προγράμματα, τα οποία έχουν στο στόχο να γίνουν πιο συγκεκριμένα κατά επόμενα έτη και βεβαίως θα αφορούν τα προγράμματα αυτά τους επόμενους 18 μήνες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα βρίσκεται μπροστά σε πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία η οποία θα πρέπει κάποτε να παρουσιάσει ανάπτυξη μετά από όλα αυτά τα χρόνια της ύφεσης. Η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι οι πρώτες προτεραιότητες της Προεδρίας μας και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να υιοθετήσουμε στρατηγικές οι οποίες θα επιτρέψουν στην ενέργεια να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα περάσω τώρα με λεπτομέρειες στις προτεραιότητες ε, του εξαμήνου μας κατά, στους τομείς ενέργεια και ε, ανταγωνιστικότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε στο Συμβούλιο σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων ε, και προστίθεται βέβαια και η κρίση η Ουκρανική, άρα δηλαδή πρέπει ακόμα πιο στεναρά να διεκδικήσουμε τους στόχους μας που είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η ενεργειακή ασφάλεια, η πλήρης ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών. Όσον αφορά το νομοθετικό έργο, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μαζί με το Κοινοβούλιο έχουμε ε, καταλήξει σε ένα σημαντικό ε, χαρτοφυλάκιο, ένα νομοθετικό έργο, την ε, οδηγία iLook. Από την ελληνική προεδρία, η δική μας η προεδρία είναι πρόθυμη να ξεκινήσει τον άτυπο διάλογο με τους αρμόδιους ευρωβουλευτές. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές προτεραιότητες, είμαστε υπέρ του να υπάρξει μια συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου όσον αφορά το θέμα πλαίσιο για την ενέργεια και για το ε, και τις αλλαγές. Αρμόδια βέβαια για αυτά τα θέματα είναι και ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, οι Επιτροπές και τα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας. Στις 6 Οκτωβρίου στο Μιλάνο θα γίνει μια σχετική συνάντηση. Θα υπάρξει πρώτη ανταλλαγή απόψεων, κυρίως όσον αφορά την ανακοίνωση Επιτροπής για την ενεργειακή ε, επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Αυτή έγινε στις 23 Ιουλίου και αναφέρει ότι θα πρέπει να, περιοριστούν, ε, να περιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά 30% μέχρι το 2030. Υπάρχει και το σχετικό πακέτο πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα είναι μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά του ε, φιλόδοξους στόχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την προηγούμενη θητεία. Η εξοικονόμηση τη ενέργεια από κοινού με τις ανώσιμε πηγές ενέργειας είναι ένα στοιχείο κλειδί που μπορούν να βοηθήσουν στο να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η ε, δέσμευσή μα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων δεν σημαίνει ότι έχουμε ε, μία μαγική συνταγή για όλου. Θα πρέπει να δούμε τι εθνικέ ιδιαιτερότητε, την τεχνολογική ουδετερότητα και όλα αυτά έχοντας κατά νου τις επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν σε άλλους τομείς, κυρίως στη βιομηχανία και στην εργασία. Εμείς λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή προσέγγιση και θέλουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να βρούμε μια στρατηγική η οποία θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ακολουθήσει αυτόν τον φιλόδοξο δρόμο της απεξάρτησης από τον άνθρακα. Έχουμε διεθνείς ε, κρίσεις ε, και αυτή της Λιβύης και της Ουκρανίας και αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια εντελεχή μελέτη όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και αυτό θα ξεκινήσει ε, σύντομα μετά από την συνάντηση των G7 που έλαβε χώρα στο, στη Ρώμη τον Μάιο. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τον ενεργειακό εφοδιασμό και αυτοί αφορούν τις εξελίξεις στη Ρουσία και στην Ευρώπη. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου η Ιταλική Προεδρία έχει διδρομολογήσει συζήτηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια μέσω μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτηση που αφορούν τους υπουργού Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποβληθούν επιβληθούν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και η ενεργειακή επάρκεια θεωρούμε ότι θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να απεξαρτηθεί από ενεργειακούς πόρους. Το αέριο θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση προς ε, την απεξάρτηση από τον άνθρακα και βέβαια ε, η προμήθεια, η εφοδιασμός με άνθρακα για την Ευρώπη είναι σήμερα απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αξιολογήσουμε και την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής, να καταλήξουμε σε ουσιαστικές σχέσεις με τους προμηθευτές. Εν τω μεταξύ είναι απαραίτητο να υλοποιήσουμε τις πιο σημαντικές υποδομές που αφορούν κυρίως το άνοιγμα του ε, διαδρόμου προς νότον και την σημασία που πρέπει να αποδώσουμε στο υγροποιημένο αέριο. Είναι πράγματι σημαντικό να υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες υγροποιημένου αερίου. Η Ιταλική Προεδρία και Επιτροπή συμφώνησαν στο να ξεκινήσουν κυρίως ε, σχέσεις και διαπραγματεύσεις για τα ευρωμεσογειακά θέματα. Στις 19 Νοεμβρίου στη Ρώμη θα υπάρξει και άλλη μια συζήτηση για, το ευρω... για την ευρωμεσογειακή ενεργειακή σχέση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακαλούμε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και το πώς μπορεί η Αφρική να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια. Οι προσπάθειε μας για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, οι προσπάθειες αυτές ε, είναι ε, μερικές θα έλεγα για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Μετά το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2011 σκοπεύουμε να προτείνουμε ένα κείμενο και συμπεράσματα που αφορούν στο τι υπολείπεται ακόμα για να γίνει. Επίσης τα συμπεράσματα αφορούν την ε, ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελπίζουμε να λάβει χώρα σύντομα. Στην θητεία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα ακολουθήσουν ε, προτάσεις που βασίζονται στη δουλειά που έχει γίνει για τη σημασία της ενέργειας. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να συμμετέχουν και οι ε, καταναλωτές μέσα από την διάχυση εφιών τεχνολογιών. Στο Συμβούλιο πρέπει να εντοπίσουμε το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν όπως η ολοκλήρωση της κοινή αγοράς. Αυτό αφορά το πλαίσιο για θέματα υποδομής αλλά και για θέματα που είναι διασυνοριακά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα διασύνδεσης και του αποκαλούμενου reverse flow. Επίσης να κάνουμε χρήση του κανονισμού για τα ενεργειακά ευρωπαϊκά δίκτυα. Η Ευρώπη ε, χρειάζεται 5 δισεκατομμύρια επιπλέον για τις ενεργειακές υποδομές ε, κατά τα επόμενα 7 έτη. Για να έχουμε τα 200 δισεκατομμύρια το συνολικό ποσό που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις επενδύσεις στον τομέα. Πρέπει να γίνουν μελέτες περαιτέρω τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε να εφαρμόζονται πλήρως οι κανονισμοί στην κοινή αγορά, να αυξηθούν οι διασυνοριακές ανταλλαγές στον τομέα της ενέργειας, να υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης, επιθυμούμε τα αποτελέσματα που υπάρχουν ήδη να οδηγήσουν σε μια πιο στενή περιφερειακή συνεργασία. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες του προγράμματος της Προεδρίας όσον αφορά την βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη που βασίζονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου και του Ιουνίου. Τα βασικά, βασικοί στόχοι αφορούν ε, τις δραστηριότητες που αυτό ε, αναπτύξαμε και σκοπεύουμε να αναπτύξουμε κυρίως όσον αφορά την governance στον βιομηχανικό τομέα και την ολοκλήρωση της βιομηχανικής πολιτικής σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το mainstreaming. Αυτά τα δύο θέματα τα εξετάσαμε ήδη τον Ιούλιο μετά την ε, άτυπη ή κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών στο Μιλάνο και εκεί επιτεύχθηκαν τρία σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν σε πολιτικούς στόχους, στην ενίσχυση της governance και στην ε, βιομηχανική πολιτική και στη ε, διάσταση της πολιτικής αυτής που πρέπει να παρισφρήσει σε πολλές άλλες. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη δημιουργία υπεραξίας στο βιομηχανικό τομέα της τάξης του 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Η Προεδρία προάγει συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου για να συμβάλλουμε και εμείς στην αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και για να συμπεριληφθούν οι στόχοι της αναθεώρησης σε έναν ευρύτερο πλαίσιο. Στο Μιλάνο προέκυψε ευρεία συνένεση ε, και συμφωνία των Υπουργών ε, στο να συσταθεί ένα, μια ομάδα υψηλού επίπεδου, αλλά αυτή η ομάδα να μετατραπεί τελικά σε μια σταθερή ομάδα με μόνιμη προεδρία και να εργάζεται τουλάχιστον για 18 μήνες. Εμείς θα συμβάλλουμε στο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ένα άλλο στόχο που σας ανέφερα, δηλαδή το στόχο του mainstreaming αυτής της διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής, αυτό αφορά τις ε, βιομηχανικές πρώτες προτεραιότητες. Θεωρούμε ότι αυτές είναι το κλειδί για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ήδη λοιπόν στο Μιλάνο ε, αναφέρθηκαν διάφορες παραδοχές. Σκεφτήκαμε να υπάρχει και μια τομεακή προσέγγιση η οποία ε, θα επιτρέψει να υλοποιηθεί το mainstreaming σε ορισμένους τομείς ε, κατά τα επόμενα δύο έτη. Και αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπάρχει μία βάση έτσι ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε την απαραίτητη μέθοδο ακόμα και σε πολύ περίπλοκους τομείς. Το Συμβούλιο του Μιλάνου επιτεύχθηκε ε, σχεδόν ομοφωνία όσον αφορά τις επιπτώσεις της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία από τις πρόσφατες πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα του υψηλού κόστους της ενέργειας και της ύπαρξης ενεργοβόρων βιομηχανιών σε διάφορους τομείς. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει και αυτή ότι πράγματι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν, γι' αυτό υπάρχει και το Fitness Check και το πρόγραμμα Refit. Ήδη έχει υπάρξει αξιολόγηση σε ορισμένους τομείς, ο έλεγχος της ανταγωνιστικότητας πρόκειται να λάβει χώρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της εφιούς ρύθμισης. Η Ιταλική Προεδρία επιθυμεί οι στόχοι και ο χάρτης πορείας να περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου ανταυτού μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για να υιοθετήσουμε γενικότερα συμπεράσματα για τη βιομηχανική πολιτική ακόμα και κάτω από το πρίσμα των προτεραιοτήτων και των στόχων του στρατηγικού θεματολογίου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες προτεραιότητες του προγράμματος της Προεδρίας είναι οι πολιτικές προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο Συμβούλιο το Δεκέμβρη προβλέπεται για πρώτη φορά η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως των envoys των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά στην υλοποίηση του Small Business Act. Εμείς θέλουμε να προάγουμε τον πολιτικό διάλογο για το Small Business Act, ε, κυρίως ε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι το 2015. Η Ιταλική Προεδρία επιθυμεί να ευνοήσει την υλοποίηση ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη της ε, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του παραγωγικού συστήματος, Θέλουμε να έχουμε παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στο να προβάλλεται η μικρή διάσταση, να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια της, στην ανάπτυξη όπου υπάρχουν αυτά και επιθυμούμε επίσης, επιθυμούμε να φέρουμε ισορροπία σε διάφορους ε, παράγοντες που οδηγούν ε, σε μείωση της παραγωγής. Πριν ολοκληρώσω θέλω να σας πω ότι η Προεδρία μας ε, θα φιλοξενήσει το Νοέμβρη, στην, θα φιλοξενήσει στην Νάπολη την τρίτη ετήσια συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, μία συνάντηση όπου τα συμμετέχουν πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρους. Πάνω από 500 μετέχοντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήματα που έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Μια ενέργεια Όντω είναι πολύ σημαντικό θέμα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Βέβαια, υπάρχει και σφαιράρι που είναι ιταλική μάρκα σήμερα. Αλλάζουμε όμως θέμα τώρα και περνάμε στις τηλεπικοινωνίες. Αντωνέλο Τσακομέλη, υφυπουργός αρμόδιος για τις τηλεπικοινωνίες. Δημοσιογράφος με μεγάλη εμπειρία και εκδότης. Αλλά και στην αυτοδιακυβέρνηση, γιατί ήταν δήμαρχος και ενίσχυσε πολύ τις τοπικές υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα της ενέργειας και των δικτύων. Να, η αρχή της ε, δικιάς σας συμμετοχής στην Ιταλική κυβέρνηση. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιδήμαρχος ήμουνα στο πράγμα, όχι δήμαρχος, αλλά ευχαριστώ πάντως που με ανεβάσατε. Ευχαριστώ και για την διάθεση που δείξατε να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τις απόψεις της Ιταλικής Προεδρίας για τις ε, προτεραιότητες που θέλουμε να προωθήσουμε σε αυτόν τον τομέα κατά τη διάρκεια των, του εξαμήνου μας. Η ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτικής έχει στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη, την απασχόληση στην Ευρώπη και για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έδειξε αυτό με μια πρόσφατη έκθεση που εντόπισε την πλήρη απουσία της ε, ψηφιακής πολιτικής ε, ενιαίας αγοράς ένα από τα βασικά προβλήματα τη της Ευρώπη. Ευρώπης. Ο πρόεδρος Γιούνκερ άλλωστε στο πρόγραμμά του υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ψηφιακής αγοράς που θα έδινε ανάπτυξη κατά 500 δις μέχρι το 2020 προς ε, όφελος των πολιτών και των χωρών. Η ιδέα λοιπόν της υλοποίησης ε, της ε, ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς είναι αυτή που θα οδηγεί τη δουλειά μας. Ακόμη περισσότερο δε μας παροτρύνει η φιλοδοξία να κάνουμε την Ευρώπη το είπε ο Πρωθυπουργό κ. Ρέντσι στο παρελθόν στην εκδήλωση στην Βενετία του Digital Venice. Στόχος μας είναι να κάνουμε την Ευρώπη ένα πολιτικό και θεσμικό υποκείμενο ικανό να διαμορφώσει κοινέ ψηφιακές πολιτικές. Η Ιταλική Προεδρία για το σκοπό αυτό θα παίξει το ρόλο της παροχής διευκόλυνσης και συμβολής από τις απόψεις των διαφόρων κοινωνικών κυβερνήσεων. Τρία είναι τα βασικά θέματα επί των οποίων δουλεύουμε η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ασφάλεια και το web, το δηλαδή, και το web accessibility, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Για την ψηφιακή ενιαία αγορά βεβαίως το θέμα προτεραιότητας, το net neutrality, η ουδετερότητα του δικτύου είναι ένα θέμα που είχε σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το ξεκίνημά του μετά την απόφαση ιδίω του Federal Communication Commission τον ΗΠΑ που άνοιξε το δρόμο για κάτι που διαπιστώνεται όλο ένα και περισσότερο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και των λεγόμενων over the top. Είναι σημαντικό ότι ε, αν τόσο ο δρόμος ακολουθεί θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέπει να συνδέει την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου με την ισότητα πρόσβασης και ευκαιριών στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μην υπάρξει μόνο μία εμπορική διάσταση της προσέγγισης αυτής, αλλά τα θεσμικά όργανα και η ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων σε εθνικό επίπεδο θα είναι καλύτεροι να προστατεύσουν το δίκτυο όπως το γνωρίζουμε, ως ένα χώρο δηλαδή ευκαιριών και ελευθερίας, ως ένα χώρο ενιαίο, μοναδικό, μη διαιρούμενο, ικανό να εξασφαλίσει ασφάλεια και στην έκφραση του καθενός και την παροχή εμπορικών δυνατοτήτων, ε, ε, ε, δυνατοτήτων εμπορικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να αποφευχθεί ωστόσο συμφωνίες μεταξύ γιγάντων του εμπορικού κόσμου που ενδεχομένα δημιουργήσουν εμπόδια στην είσοδο στο δίκτυο παρεμποδίζοντας τη δυνατότητα νέων να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ. Το roaming είναι το άλλο θέμα που επικεντρώνουμε τη δουλειά μας. Το κοινοβούλιο άλλωστε έδωσε και ένα σημαντικό μήνυμα που περίμεναν πολύ. Ε, από την άποψη αυτή είναι σημαντικό να συνδυάσουμε τη δυνατότητα άρσης αυτού του εμποδίου όχι θεωρητικού αλλά και πραγματικού εμποδίου στην επικοινωνία στην Ευρώπη με τη δυνατότητα διατήρησης παρά τα αυτά κάποιες χώρες το υπογράμμισαν αυτό των επενδύσεων των εταιριών τηλεπικοινωνίας και των υποδομών τους. Η ασφάλεια είναι βεβαίως το θέμα επί του οποίου συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές μας. Από την άποψη αυτή, στο τελευταίο Συμβούλιο έγινε μια σημαντική συζήτηση με συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες θέσεις των διαφόρων κυβερνήσεων. Υπάρχει κοινή επίγνωση της ανάγκης να υπάρξει ένα αποφασιστικό και ενιαίο βήμα προς τα μπρος από πλευράς Ευρώπης στο ζήτημα αυτό. Υπάρχει μια διαθεσιμότητα εν γέννη για, για στρατηγική συνεργασία, ούτως ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για μια συνεργατική προσέγγιση, βαθμιαία ενδεχόμενα, για να υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση δίπλα στα θέματα αυτά. Εμείς από πλευράς μας θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διακυβέρνησης του ίντερνετ ως ένα σημείο όχι μόνο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά και πολύ, σημαντικής, ε, και πολύ σημαντικού ρόλου ε, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την Ευρώπη. Εμείς για το θέμα αυτό μάλιστα προγραμματίσαμε και ένα άτυπο συμβούλιο των τηλεπικοινωνιών που θα γίνει στο Μιλάνο στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Πιστεύουμε ότι η εξέδειξη του ICAN είναι το τελικό σημείο για μας. Δεν θέλουμε δίκτυο κυβερνήσεων, αλλά ένα δίκτυο που οι χρήστε θα είναι πρωταγωνιστέ και θα έχουν δυνατότητε ελευθερία και ευκαιριών. Πιστεύουμε ωστόσο ότι πρέπει να δουλέψουμε μετά την αλλαγή των θέσεων των ΗΠΑ προ μια θετική εξέλιξη του ICAN. Και είναι θεμελιώδες κατά την άποψή μας στο ζήτημα αυτό η σχέση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ μιας Ευρώπης που είναι ικανή να αποκτήσει μια κοινή ενιαία θέση και τον είπα Αυτός είναι ο άξονας πάνω στο οποίο το δίκτυο μπορεί να εξελιχθεί και να παγιωθεί στην ανάπτυξή του. Η ευχή, βεβαίω με την οποία κλείνω την παρουσίασή μου αυτή, είναι να υπάρξει από κοινο, πλευρά Κοινοβουλίου και ιδίω Επιτροπή διαθεσιμότητα, βούληση να δεσμευθούν για μια πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τις τρεις βασικές οδηγίες που μπορεί να σηματοδοτήσουν και την επιτυχία μιας προεδρία μια ομάδα ατόμων, αλλά ταυτόχρονα και ακόμη περισσότερο ένα μήνυμα τη ικανότητα τη Ευρώπη ότι θέλει και μπορεί να είναι ένα πολιτικό υποκείμενο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Προχωρούμε στις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Τρία λεπτά μάξιμου ανά συντονιστή. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, εκτιμήσαμε την θέση της Ιταλικής Προεδρίας, ιδίω διότι και τη δουλειά που κάνει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2014 που δημιούργησε αυτό το Industrial Compact και που έλαβε πολλές θετικές ε, πολύ θετική υποστήριξη, τουλάχιστον στην, στη Σύνοδο Κορυφή του ΕΛΚ. Εμεί ε, θεωρούμε ότι το να υπάρξει μια πραγματική βιομηχανική πολιτική τη Ένωση που θα μα επιτρέψει να φτάσουμε στο στόχο μα είναι κάτι σημαντικό. Βεβαίω το θέμα τη ενέργεια, όπω υπογραμμίσατε, ε, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να έχουμε βιομηχανική πολιτική αν δεν υπάρχει μια προσπάθεια μείωσης του κόστου ενέργειας που λόγω της οικονομική κρίσης κινδυνεύει να αυξηθεί. Πόσο μάλλον που με την κρίση στη Βόρεια Αφρική, την Λιβύη ιδίω ε, επιδεινώνεται. Πρέπει λοιπόν να λυθεί γρήγορα η διαφορά που εμφανίζεται εκεί. Νομίζω ότι είναι θετική η δράση και της Ιταλικής κυβέρνησης ως προεδρευούσης να αντιμετωπίσει το θέμα του carbon leakage. Ε, είναι σαφές ότι η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται μία προσεκτική δράση στη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος με στόχους επιτεύξιμους και όχι με στόχους που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Συμφωνώ επίσης με όσα είπατε, με όσα είπε ο κ. Τζακομέλη για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενίας αγοράς, που είναι ένα εργαλείο ανταγωνιστικότητας και επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασία ποιότητα. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ωστόσο και την ανταγωνιστικότητα τη ψηφιακή αγορά, προσφέροντα ε, και δυνατότητε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μπροστά στην είσοδο στην αγορά γιγάντων, ε, γιγαντιαίων επιχειρήσεων από τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία. Πρέπει να προστατεύσουμε και τη βιομηχανία τη Ευρώπη με ένα σύστημα level playing field. Είναι σημαντικό επίση και αυτό που είπε και ο Υπουργό, να δουλέψουμε ούτω ώστε να υπάρξει ένα screening για κάθε το ζήτησε η Επιτροπή, νομοθετική απόφαση που έχει θετικέ ε, δηλαδή τίθεται στην βιομηχανική πολιτική. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό, να δώσουμε δηλαδή στο Συμβούλιο αντιγωνιστικοτητα μεγαλύτερε εξουσίε. και ελπίζω η, προεδρία, η Ιταλική Προεδρία να δώσει ζωή σε, αυτή, σε αυτό το Συμβούλιο Βιομηχανία που θα είναι το άλλο, ο άλλο πυλώνα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Ένα σημείο κατά την άποψή μου λείπει στι παρεμβάσει η πρόσβαση στην καταναλωτική πίστη των μικρομεσαίων κυρίω επιχειρήσεων. Χρειάζεται ισχυρότερη δράση από πλευρά Συμβουλίου. Είδαμε βέβαια ότι ο προπολογισμό του 2015 τουλάχιστον στις προτάσει του Συμβουλίου, περικόπηκε ιδίως σε κάποια σημεία που αφορούν την βιομηχανική πολιτική, την πολιτική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα η Επιτροπή υπερψήφισε την αποκατάσταση του προϋπολογισμού Ιδίω τι χρηματοδοτήσει για τι επιχειρήσει και την πραγματική οικονομία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα χτυπήσουμε την κρίση και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ει βάρο τη πραγματική οικονομία των παραγωγών αυτών που δίνουν θέσει εργασία. Γι' αυτό ζητούμε παρέμβαση από πλευρά τη Ιταλική Προεδρία, δυνατή παρέμβαση για να αποκατασταθεί ο προπολογισμό όπω ήταν. Κλείνω, Πρόεδρε χωρίς βιομηχανία, χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την κοινωνική οικονομία αγοράς που όλοι θέλουμε και επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόγια, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ιταλικής Προεδρίας για την παρουσία τους εδώ και αυτά που μας είπαν αλλά και για τη δουλειά που θα κάνουν του επόμενου τους μήνες. Και βεβαίως ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστούμε επίσης ε, και για την διαθεσιμότητα που δείχνουν. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι θέλουν να συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια ε, της, ε, του συνόλου της ε, Προεδρίας. Πράγματι πρέπει να υπάρχουν πιο ισχυρές πολιτικές σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτά που είπε ο κ. Γκουίντι γιατί για τα άλλα θέματα θα τεθούν αυτά από τους συντονιστές και από άλλους Ιταλούς Ευρωβουλευτές. Αυτά που μας είπατε πράγματι απασχολούν την Επιτροπή μας και συμφωνούν συμφωνούμε απόλυτα με αυτά. Όλοι μας θέλουμε η πολιτική, η βιομηχανική να εξελιχθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχυθεί η governance. Ε, η έννοια, η ιδέα ενός ε, Συμβουλίου Υπουργών Βιομηχανίας είναι κάτι που το προάγουμε εδώ και πολύ καιρό. Γιατί στην, ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας η βιομηχανική πολιτική είναι απλά μία διάσταση. Όμως ο στόχος τελικά είναι να υπάρχει μία ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Και αυτά που είπατε για τις ομάδες υψηλού επίπεδου, για το mainstreaming, αυτή η πολιτική ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναθεωρηθεί. Γιατί δεν είναι ανταγωνισμός που επιτρέπει την ανάπτυξη, αλλά είναι μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική που πρέπει να έχει περισσότερο σχέση με την ανταγωνιστικότητα προς τα έξω. Ε, κάποια θέματα που έχουν σχέση, παραδείγματο χάρη με το χάλιβα και άλλα, αντιμετωπίστηκαν ε, κατά το παρελθόν με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε επ' αυτών. Και θέλω να πω κάτι σχετικά με το 20% του ΑΕΠ από τη βιομηχανία. Η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια ε, επιδίωξε κοινού στόχου, αλλά όσον αφορά τα εργαλεία πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία. Ε, πράγματι δέχομαι ότι θα πρέπει να μπει κανεί κάνει στην ουσία των θεμάτων λίγα λόγια και συγκεκριμένα εργαλεία. Το θέμα των επενδύσεων, ε, το θέμα της ανταγωνιστικότητα. Σήμερα ακούσα μια σχετική μελέτη. Η πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια ε, θα πρέπει λοιπόν να πει κάποιος ε, στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους αρμόδιους ότι τα δάνεια πρέπει να δίδονται στη βιομηχανία. Και ποιος θα το κάνει αυτό, οι επενδύσεις ε, για φέτος ε, δεν προβλέπονται πολλές κρατικές επενδύσεις και πώς θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. Να υπάρξουν κρατικές επενδύσεις στην έρευνα, παραδείγματος χάρη. Φοβόμαστε λοιπόν να μιλάμε για αυτά τα θέματα, αλλά τώρα λοιπόν το Συμβούλιο ε, μπορεί κάτι να κάνει και θέλω να προσθέσω και ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Θα ήθελα να προσθέσω και το θέμα των εργαλείων ε, που είναι στοιχεία μόχλευσης, ε, οι εγγύησει, το sharing risk ε, και τα παρεμφερή. Με την Ιταλική Προεδρία μπορούμε να συζητήσουμε και για τον επόμενο προϋπολογισμό έτσι ώστε να δραστηριοποιήσουμε, να δραστηριοποιήσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο. Ξεκινώντας βέβαια από το κρατικό κεφάλαιο έρευνα και τεχνολογία δεν γίνεται αρκετή χρήση των αποτελεσμάτων. Η Ιταλική λοιπόν Προεδρία μπορεί επ' αυτών ε, να προχωρήσει έτσι ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει και στο θέμα αν θέλετε του προγράμματος Horizon. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε, εδώ να κάνουμε την αρχή. Ξέρω ότι έχω καθυστερήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τόγια. Τώρα, στη συνέχεια κύριος Κρομπάρτσιφ από τους Ευρωπαίους Διευθυντικούς. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στη γλώσσα μου. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι Υπουργοί, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τις τόσο πλήρης παρουσιάσεις σας. Θέλω να σας ευχηθώ επίσης κάθε επιτυχία στο έργο σας. αναφερθήκατε στην επίτευξη των στόχων της ατζέντα για το 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν τον άθρακα πλήρως, τι θα χρησιμοποιήσουμε λιβικό αέριο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην τεράστια αστάθεια που επικρατεί σε χώρες όπως αυτή και σε διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό όμως γιατί όπου να είναι θα έχουμε χειμώνα στην Ευρώπη. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε, να επιλέξουμε λιβικό ή γενικότερα να το πω αφρικανικό αέριο για να ανταποκριθούμε στις ενεργειακές μας ανάγκες. Και πώς. Η οικονομία μας σήμερα δεν είναι ανταγωνιστική απέναντι στην Αμερική. Συνεπώς, πώς και πότε θα έχουμε ανταγωνιστικότητα και θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιες λύσεις όπως είναι το αφρικανικό αέριο. Όταν θα έχουμε ανταγωνιστικότητα λοιπόν χρησιμοποιώντας αυτό το αέριο, τι θα κάνουμε μετά με το σχιστολιθικό αέριο. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού και σχετικά με την ρογμάτωση. Πώς βλέπετε τις προοπτικές εκμετάλλευσης του συστολιθικού αερίου. Πόσο σημαντικό είναι για σας αυτό το θέμα, το θεωρείτε σημαντικό ή όχι. Στην ε, ψηφιακή αγορά τώρα. Αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων την διαχείριση του διαδικτύου. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχαμε να εξετάσουμε την άκτα. Πολύ επίμαχο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Για πείτε μας λοιπόν παρακαλώ. Πώς θα δράσετε εσείς όσον αφορά τη διαχείριση του διαδικτύου. Πρόεδρος. Ο κύριος Πέτερσεν είναι ο επόμενος ομιλητής, επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, εκ μέρους της Άλντε. Παρακαλώ κύριε Πέτερσεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε σήμερα με την Ιταλική Προεδρία. Με πολύ χαρά άκουσα τις παρατηρήσεις σας και για την ε, διακυβέρνηση, για τη διαχείριση του διαδικτύου, για την περιαγωγή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε υπόψη ότι το διαδίκτυο φτιάχτηκε σαν μια ανοιχτή πλατφόρμα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το διατηρήσουμε ως ανοιχτή πλατφόρμα. Οπότε συγχαρητήρια για αυτά που μας είπατε και μην ξεχνάμε αυτόν τον αγώνα προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το διαδίκτυο. Οι ερωτήσεις μου τώρα έχουν να κάνουν περισσότερο με την ενέργεια. Άκουσα να λέτε πολλά καλά για την ανάγκη να χρησιμοποιούμε περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση επίσης. Αλλά θα ήθελα να γίνετε πιο συγκεκριμένοι. Τι σημαίνει αυτό, τι χρειάζεται για να γίνει αυτό, ποιοι θα είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι που θα ζητήσετε στις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα. Θα πιέσετε για πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια ή για την ε, ενεργειακή απόδοση. Ξέρω ότι είναι δύσκολη δουλειά, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό εμείς να σχηματίσουμε μια πραγματική εντύπωση για το πού θέλει να μας οδηγήσει η Ιταλική Προεδρία. Σας ευχαριστώ και πάλι για τόσα μας είπατε. Πρόεδρος και εμείς. Ευχαριστούμε κυρία Λόπες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, της ΓΟΕ. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Θέσατε φιλόδοξους στόχους, όμως η πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται έχει πάρει άλλο δρόμο. Θα είναι δύσκολο να πετύχουμε έτσι κι αλλιώς το στόχο του 20% του, του... του ΑΕΠ για την βιομηχανία. Τη στιγμή που έχουμε δει ότι σε αυτή την περίοδο κρίσης το ΑΕΠ έχει μειωθεί και ότι τα κονδύλια τα οποία πηγαίνουν για επαναβιομηχανοποίηση δεν επαρκούν. Το είδαμε αυτό πόσο ανεπαρκής είναι η χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού για επαναβιομηχανοποίηση. Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες γίνεται το αντίθετο. Υπάρχει μια πολιτική από βιομηχάνωσης και όχι το αντίθετο και όχι ενίσχυση τη βιομηχανία. Χρειάζονται λοιπόν επενδύσει στις υποδομέ σίγουρα. Χρειάζονται όμω επενδύσει από το δημόσιο δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλο είδου επενδύσει. Ο δημόσιο τομέα είναι εκείνο ο οποίο πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση και να δώσει επενδύσει. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν έχει αναφερθεί και μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα της δικιάς μας Επιτροπής αλλά είναι ευρωπαϊκό θέμα και αυτό είναι η φορολογική εναρμόνιση προκειμένου να ισχύουν οι ίδιοι όροι για όλε τι επιχειρήσει, Γιατί αλλιώ, ο στόχος της ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν θα επιτευχθεί εύκολα, για να μην πω καθόλου. Εκτός αν οι θέσει απασχόλησης που δημιουργούνται, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, είναι θέσεις που ανταποκρίνονται σε ανθρώπους με ελάχιστα προσόντα και με πολύ χαμηλούς μισθούς που οδηγούν σε φτώχεια και ανισότητα τους πολίτες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και την εγκατάλειψη του άνθρακος, έχω να σας πω το εξής. Υπάρχει η Ενάγας που είναι μια ισπανική εταιρεία, μια επιχείρηση που δημιουργήθηκε με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία και παίρνει τα πόβλητα από τον άνθρακα και τα κάνει ενέργεια πρόκειται να κλείσει. Θα κλείσει το Δεκέμβριο, διότι η Ισπανική κυβέρνηση είπε ότι οι ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας δεν είναι προτεραιότητα. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρώπη ώστε οι χώρες να βάλουν ως προτεραιότητα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να το τηρήσουν αυτό. Οι επιχειρήσεις λοιπόν σαν κι αυτήν είναι αυτές τις οποίες πρέπει να στοιχηματίζουμε όπως και η Ευρώπη υψηλή ποιότητας με ανθρώπους που έχουν τις σωστές δεξιοτεχνίες που είναι αηφόρες επιχειρήσεις υπέρ των ανανόσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή μας λοιπόν αλλά και η Προεδρία τους επόμενους 18 μήνες μια που έτσι καλώς οι Προεδρίες συνεργάζονται μεταξύ τους, θα ήταν πολύ θετικό να λάβουν υπόψη τους την πρόταση αυτή για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης και αυτά τα οποία λένε τα συνδικάτα που λένε ότι μπορούν να, να υπάρξουν ε, πάρα πολλές νέες θέσεις απασχόλησης αν έχουμε έναν καλό σχεδιασμό για την επαναβιομηχανοποίηση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έριξον τώρα, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος και τους δύο μας ομιλητές. Σας ευχαριστούμε που μας θέσατε τις προτεραιότητές σας. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι θα ήταν Καλύτερα μάλιστα αν μας δείχνατε συγκεκριμένα βήματα που θέλετε να αναλάβετε στους τομείς αυτούς. Γιατί αυτό μας απασχολεί στην Ευρώπη. Να ξέρουμε τι βήματα θέλετε να γίνουν για να δούμε και εμείς πώς θα τα κάνουμε και πώς θα βοηθηθεί, θα βοηθήσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες μέλη για να βελτιώσουν το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας να ενισχύσουν ε, τις, ε, τη χρήση των ε, εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Και θα έλεγα και ένα πράγμα ακόμα. Θα ήθελα κι εγώ, σαν προτεραιότητα, κάτι κατά της διαφθοράς. Όντω στην Ευρώπη αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια αν θέλουμε καλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η Ιταλία, για παράδειγμα, πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλή θέση για να μας δείξει πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Δάριο Ταμπουράνο τώρα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την πολύ ωραία παρέμβασή σα, Ό,τι αφορά όμως τη στρατηγική ασφάλεια ενέργεια τη ε, Ένωση, 31 Ιουλίου στην Ιταλία με την κυβέρνησή σα η, μια κινέζικη επιχείρηση πήρε το 35% του CDP rating που αγοράστηκε και απονομίζεται State, State Corporation of China η ιδιοκτησία της κινέζικης ε, κυβέρνησης που ελέγχει το 35% των αποθεματικών αερίου και κατά συνέπεια έχουν δυνατότητες παρέμβασης όχι μόνο στα δίκτυα αλλά και στη διασύνδεση μέσω Ιταλίας μεταξύ των ε, της βορείου, του αερίου της, βορείους, ε, της Βορείου Αφρικής και της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Καθώς η, η παρέ, όπως γινόταν και στην πρώτη κυβέρνηση και στην πρώτη δημοκρατία της Ιταλίας, όλα αυτά έγιναν καλοκαίρι χωρίς να ξέρει τίποτα ο πολίτης. Δισεκατομμύρια ε, μετακινήθηκαν. Αυτό είναι, πολιτικές, είναι οι συνέπειες της πολιτικής λιτότητας που υποχρεώζουν, υποχρεώνουν τα κράτη της Ένωσης να μαζεύουν χρήματα από παντού εις βάρος της μακροπρόθεσμης προοπτικής των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, το ότι αυτή τη στιγμή κομμάτι της Ιταλίας ανήκει σε εξοκοινωτική κυβέρνηση, τι, απο, τι, τι σας κάνει να πιστεύετε, πώς αξιολογεί η ίδια η Επιτροπή την εξέλιξη αυτή. Να προσθέσω σε ό,τι αφορά την μετάβαση προς την ε, ε, ανανεώσιμη ενέργεια ότι η κυβέρνηση Ρέντσι οθέτησε ένα ε, διάταγμα που λέγεται Σμπλοκ Ιτάλια που διαλύει ολόκληρη την φωτοβολταϊκή πολιτική της Ιταλίας ε, πηγαίνοντας, μεταβιβάζοντας σε πολύ, μακροχρόνια, πολύ πιο μακροχρόνια περίοδο την ε, τη μετάβαση προς το βολταϊκό. Με τον τρόπο αυτό, στην ουσία, ανατράπηκε ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός επιχειρήσεων Ιταλικών και Ευρωπαϊκών, αλλά και οικογενειών. Πώς συνδυάζετε αυτές τις φορολογικές επιλογές σας με τους στόχους της Ένωσης για την ε, ασφάλεια ενέργεια και με αυτή τη δεσμεύση που περιλαμβάνουν στο πακέτο για την, για την προστασία ε, του περιβάλλοντος μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ. Παρακαλώ να απαντήσετε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων που ακούστηκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ελπίζω με κάποιο σύντομο τρόπο. Στον κύριο Ταγιάννη θέλω να πω ότι προφανώς και συμφωνώ μαζί σας. Εμείς ως Προεδρία θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τις ε, προτάσεις του Συμβουλίου του Μαρτίου για το Industrial Compact. Όσον αφορά το στόχο του 20% θέλω να σας πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να αναζητάμε το διάλογο ε, σχετικά με ένα στόχο που προφανώς ε, θα πρέπει να παραμείνει ένας ε, στόχος όχι δεσμευτικός, αλλά κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να επιδιώξουν. Δηλαδή ένας ε, στόχος ε, πολιτικά σημαντικός. Επ' αυτού βέβαια ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της ευαισθητοποίησης που δυστυχώς δεν είναι παντού ίδια. Όσον αφορά με πάση περιπτώσει την Προεδρία, το 20% είναι μια πρόταση με την οποία εμείς συμφωνούμε. Κατά τα άλλα, όσον αφορά ε, στην απεξάρτηση από τον άνθρακα και τους ενεργειακούς ε, διαδρόμους. Εμείς ως Προεδρία θεωρούμε ότι είναι κοινή στόχη, δηλαδή το 40% και το 27% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως ε, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει μία πρόταση σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια που αναφέρεται σε αυτό το στόχο, το στόχο του 30%. Και πιστεύω ότι ε, προφανώς και εμείς ως Προεδρία συμφωνούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μία καλή διαπραγμάτευση για αυτούς που είναι ήδη τρεις ε, πολύ σημαντικοί στόχοι. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει και εκείνη προτάσεις όσον αφορά τους τομείς που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην ανταγωνιστικότητα. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η δική τους η συνεισφορά σχετικά με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, το carbon leakage. Γιατί αυτό αφορά κυρίως επιχειρήσεις ε, που είναι εκτεθειμένες στην ανταγωνιστικότητα. Όσον αφορά τώρα ε, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Προεδρία γιατί κατά κάποιον τρόπο αυτή δρομολόγησε όλη αυτή τη δουλειά. Εμεί ε, είχαμε ένα άτυπο συμβούλιο στο Μιλάνο και εκεί προέκυψε σύγκληση απόψεων για το ότι είναι απαραίτητο να προάγουμε την governance στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Εμείς λοιπόν θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως θα αναζητήσουμε την ε, ενίσχυση αυτού του, ε, της ομάδας, αυτής της ομάδας υψηλού επίπουδου. Αυτό ως ένα τεχνικό εργαλείο. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως θα πρέπει ε, να αλλάξει όλη η στάση σχετικά με το mainstreaming. Υπάρχουν πολλά σημαντικά πακέτα όπως είναι η ενεργεία και το κλίμα και εκεί ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο μακροοικονομικής αλλά και μικροοικονομικής φύσεως. Και εσείς μιλήσατε για το στόχο του 20%. Άρα δηλαδή ε, ισχύει και αυτό που είπα και προς τον κύριο Ταγιάννη. Τώρα, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι ε, ως Προεδρείο οφείλουμε να ε, αναζητήσουμε περαιτέρω μελέτες και έρευνα για το ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά την ανάπτυξη ε, και είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα την ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν ήδη κάποια εργαλεία. Εμείς όμως ε, ως ε, Προεδρία θα αναζητήσουμε και άλλα εργαλεία τα οποία να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Ως Προεδρία οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, εγγύησεις ως πολλαπλασιαστές για τις επενδύσεις. Στην επόμενη ερώτηση που υποβλήθηκε σχετικά με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη χρήση του αερίου, σας είπα ότι η Ιταλική Προεδρία θα συνεχίσει να επιδιώκει το στόχο της ε, απεξάρτησης από τον άνθρακα. Βέβαια, σε μία μεταβατική φάση ε, η Ευρώπη είναι αναγκασμένη να καταφεύγει σε αυτόν παράλληλα με τη χρήση του αερίου. σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφές ε, ότι πρέπει να ζητήσουμε ένα μεσοπρόθεσμο στόχο που είναι η αυστηρή ενεργειακή ασφάλεια εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η δέσμευση άνθρακα. Όπως επίσης χρησιμοποιώνεται και το μηχανισμό reverse flow. Στην εισήγησή μου αναφέρθηκα στο θέμα των υποδομών και αναφέρθηκα στην ε, βελτίωση των υποδομών και του δικτύου κυρίως όσον αφορά το αέριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι καθοριστική σημασίας. Το σχιστολιτικό αέριο που αναφέρατε είναι μια επιλογή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αξιολογήσει κάθε κράτος μέλος. να δούμε τι είδου ε, γηγενή κονδύλια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να ε, βαδίσουμε και σε ε, συμφωνία και συμμόρφωση με τους κανόνες για την προσθέση του περιβάλλοντος. Άρα δηλαδή να υπάρχει ένα είδος ενεργειακό μείγμα και να υπάρχει καλύτερη χρήση, καλύτερη δυνατή χρήση κονδυλίων. Κύριε Πέτερσε, νομίζω ότι εν μέρει έχω ήδη απαντήσει όσον αφορά τους στόχους ε, των ανώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή ε, απόδοση. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, συμμεριζόμαστε τους στόχους που έχουν ήδη τεθεί και θα προσπαθήσουμε, όπως σας είπα, να προάγουμε το ποσοστό των ανανόσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρώ ότι πρέπει πράγματι να στηριχτούν και να επιδιωχθούν αυτοί οι στόχοι γιατί είναι πολύ σημαντικό ως Προεδρία να δώσουμε μία όθηση έτσι ώστε να έχουμε τελικά αποτελεσματικές ε, διαπραγματεύσεις για να διατηρηθούν αυτοί οι στόχοι που είναι τελικά ε, και προκλήσεις και όπου ε, πράγματι πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Όσον αφορά την κυρία Λόπες. Νομίζω ότι εν μέρη ήδη και σε εσά ε, σας απάντησα. Αναφέρθηκα και σε θέματα που δείξατε σε προηγούμενα σχόλια. Εσείς μιλήσετε και για, τον, ε, για τη φορολογική εναρμόνιση. Αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητες. Νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά περισσότερο τους αντέλφους από το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως, αναμφίβολα, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που έχει σχέση με τις δυνατότητες ε, ανάπτυξης ε, στην Ευρώπη. Και όσον αφορά τις ε, δημόσιες επενδύσεις, προφανώς Υπάρχουν ε, προτεραιότητες δικές μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε κατά το μέγιστο όλα αυτά τα εργαλεία που θα κρίνουμε κατάλληλα. Να στηρίξουμε λοιπόν κατά το μέγιστο, όπως σας είπα, τις ε, κρατικές, τις δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Απευθύνομαι στον κύριο Έριξον. Μιλήσαμε για την ενεργειακή ασφάλεια, για τις υποδομές, για τα τεστ κοπόσεως που μεταξύ άλλων τρέχουν τώρα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν σε αυτή την ανάλυση των ε, τεστ αντοχής όσον αφορά κυρίως ε, το θέμα του εφοδιασμού, του ενεργειακού εφοδιασμού. Νομίζω έχω απαντήσει αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε κύριε Ταμπουράνο, εσείς ε, θίξατε θέματα που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι καθαρά Ιταλικά, αφορούν εμά μόνο τους Ιταλούς. Να σας απαντήσω ως κάπου αλλού. Δεν νομίζω ότι εδώ είναι ο κατάλληλος χώρος. Και θέλω μόνο να πω ότι αυτά που έγιναν σε Ιταλικό στην Ιταλία δεν συμβαδίζει με αυτά που είπατε εσείς για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Δεν είναι όμως εδώ ο κατάλληλος ε, χώρος για να απαντήσουμε σε ε, θέματα καθαρά ιταλικού ενδιαφέροντος. Ε, θα τα πούμε ίσως κάποια άλλη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ο Υφυπουργός τώρα. Για την παρέμβαση του κύριου Ταγιάννη. οι ανησυχίες του για τις εγγύσεις προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που προσπάθησα να παρουσιάσω όταν μιλούσα για τους στόχους που θέτουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ακριβώς την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου, του net neutrality, με την ισότητα πρόσβασης και τον δίκαιο ανταγωνισμό. Εδώ υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή αφήνουμε τους πρωταγωνιστές της αγοράς να βρουν μόνοι τους αυτόνομα ένα σημείο ισορροπίας που σημαίνει ότι οι δυνατότεροι θα κερδίσουν περισσότερο ή θα υπάρχει η δυνατότητα που προσπαθούμε να πετύχουμε και ελπίζουμε πως θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο οι διεθνείς οργανισμοί για να διαμορφώσουν τους κανόνες. για την παρέμβαση Ροβάτσιτς. Σε ό,τι αφορά το Internet Governance, εμείς θέλουμε να παρεύουμε για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι της συμφωνίας που αναφέρατε. Κατά την άποψή μου, το βασικό είναι το συμφέρον των πολιτών, όχι των εταιριών ιδίως ό,τι αφορά τις, ε, παραβιάσεις του ίντερνετ ή τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των δημιουργών πάντα προς το συμφέρον του χρήστη, του, του, κάθε χρήστη πρέπει να προσανατολιζόμαστε. Απ' την άλλη πρέπει να αποφύγουμε μια υπερβολική παρίσφρηση στην ιδιωτική ζωή ή μια υπερβολική προβολή του εαυτού σου. Αλλιώς η παρέμβαση αυτή δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της προσωπικής ζωής του καθενός. Τα θέματα αυτά με πείθουν ακόμα περαιτέρω ότι το θέμα της διακυβέρνησης του ίντερνετ δεν μπορεί να αναλυθει μόνο από τη διάσταση της εμπορικής σκοπιάς αναφέρεται και στην ευθύνη και ικανότητα των ε, θεσμικών οργάνων να παρέμβουν. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μοντέλο που ανέκυψε Σαν Παόλο ...τον multi-stakeholder της, ε, γι' αυτό το λόγο και εγώ θεωρώ ότι ένα μοντέλο τύπου ICAN μπορεί να συμβάλλει στην σύνθεση των θέσεων των διαφορών κυβερνήσεων της Ένωσης. Συμφωνώ με τον κύριο Πέτρεσεν και τον ευχαριστώ για την παρέμβασή του ότι το ίντερνετ πρέπει να είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, ένας χώρος ευκαιρίας, ένας χώρος έκφρασης της ελευθερίας αλλά και ως ένας χώρος που θα δείχνει και την επαγγελματική ικανότητα. Εμείς θέλουμε ωστόσο το διαδίκτυο να μείνει μια ανοιχτή πλατφόρμα και Γι' αυτό πρέπει να είναι ισχυρότερη η δυνατότητα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων και των υποκειμένων που εμπιστεύονται το διαδίκτυο. Μόνο ένα ασφαλές, ελεύθερο και ανοιχτό διαδίκτυο μπορεί να είναι χώρος όπως θέλουμε να τον δημιουργήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Ο κύριος Μπονάντο πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προς την κυρία Υπουργό. Λέω, βοηθάμε τους μικρούς. Αν βοηθήσουμε πολλούς μικρούς, ωστόσο κάνουμε έναν γίγαντα. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη δεν βοήθησε τους μικρούς, αλλά τους μεγάλους. Είπατε ένα πρόγραμμα πιαθωμένο φιλόδοξο. Πάντα το λέγατε, το είπατε και πριν και τώρα και μετά αποτέλεσμα αποτυχία. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι άλλο. Μιλήσετε για ενεργειακή πολιτική. Έχετε μία σχέση παρά, παράλογη με τη Ρωσία. Καλό θα ήταν λοιπόν τον άλλο χειμώνα να δώσετε ε, στον ευρωπαϊκό πληθυσμό ε, εκατοντάδες χιλιάδων ε, sleeping bag για να μπορέσουν να τη βγάλουν. Μιλήσετε για την Άπολη τη συνάντηση της Νάπολης των μικρομε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ ήμουν σε μια, στην Νάπολη πολλές φορές, τον πίτσα, ωραία, είχε ωραία κουλτούρα, όμορφη θάλασσα. Ε, αλλά το να κάνεις εκεί μια συνάντηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σαν να κάνεις Σαχάρα ε, συνάντηση για ε, πίστες του σκι. Δεν είναι χώρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων η ε, Νάπολη. Μιλήστε για τις τράπεζες. Ίσως γιατί είσαστε λακέδες των τραπεζών. Το μόνο που κάνετε είναι να επιτρέπετε στις τράπεζες να, παίρνουν, να δανείζονται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 0,25% επιτόκιο και να το δίνουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με, με επιτόκιο 10-15%. Υποχρεώστε τις τράπεζες να που δανείζονται με 0,25 να δανείζουν με 3%. Έτσι βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, φοβάστε, δεν φοβάστε, ε, γιατί είστε φίλοι τους, τελειώνετε. Συγγνώμη πρόεδρε. Κλείνω πρόεδρε. Είμαι, ξε, καινούριος γι' αυτό. Ευχαριστώ και ελπίζω μεταξύ αυτών που θα πείτε να, είναι, ε, να πείτε κάτι αλήθεια γιατί αλλιώς αυτοευνοχίζεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό έχετε στη διάθεσή σας ο καθένας, γιατί έχουμε άλλους 14 που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γκιούρκ έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας εδώ για τόσα μας είπανε. Άκουσα και το ότι η Ιταλική Προεδρία θα είναι σημαντική για το θέμα αυτό. Ε, προφανώς και με την κρίση της Ουκρανίας η κεντρική Ευρώπη θα έπαιξε σημαντικό ρόλο για το θέμα της ασφάλειας ενέργειας. Είδαμε ότι μετά το 2006-2009 έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα της ενέργειας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις των δικτύων, το reverse flow για παράδειγμα και πολλά άλλα έργα για την αποθήκευση ενέργειας κλπ. Είναι αναγκαίο να έχουμε καλύτερη επένδυση σε νέες πηγές ενέργειας ωστόσο. Και ρωτώ, ποιες άλλες πηγές ενέργειας μπορούμε να λάβουμε υπόψη για τις ιδιαίτερα τροτές περιοχές της Ευρώπης, την κεντρική Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Φέντελη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε μεγάλες ευθύνες και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας αντιμετωπίζουμε πολλά και δύσκολα καθήκοντα. Θέλουμε εφοδιασμό ενέργειας παντού, θα έχουμε αντιμετωπίσουμε προκλήσεις κλιματικές, περιβάλλοντος, ενεργειακά ζητήματα με τη Ρωσία. και βέβαια παραμένει και η οικονομική κρίση. Η Ευρώπη έπειτα είναι πολύ διχασμένη. Εγώ είμαι από την ε, Σουηδία. Έχουμε έναν Υπουργό για τις επιχειρήσεις που θέλει ένα ενεργειακό σύστημα που να βασίζεται 100% στις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός είναι ο στόχος του κομματός μου και στόχος της πολιτικής συζήτησης στη Σουηδία. Τι μπορεί να κάνει η Προεδρία λοιπόν προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το χάσμα όσον αφορά το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη. Βασιζόμαστε εδώ πολύ περισσότερο σε ιδέες όπως είναι το σχιστολιθικό αέριο, χρησιμοποιούμε ακόμα άνθρακα. Παρ' όλα αυτά είναι γνωστό ότι πολλές νέες θέσεις απασχόλησης θα προέρθουν από τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάρης. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Κάρινς. Έχω μία ερώτηση. Είπατε ότι η ασφάλεια ενέργειας και η εγκατάλειψη του άνθρακα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν όμως βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα, βλέπουμε ότι πάρα πολλές χώρες, η Πολωνία για παράδειγμα, θα σήμαινε αν δεν χρησιμοποιεί τον άνθρακα η Πολωνία, ότι θα χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο. Άρα περισσότερες εισαγωγές από τη Ρωσία, που ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ ασταθές. Ή που θα έπρεπε να εισάγουμε από τη Βόρεια Αφρική αέριο. Και εκεί η κατάσταση είναι πολύ αθραυστή. Πώς θα τετραγωνίσουμε λοιπόν αυτό τον κύκλο, για να το πω έτσι. Θα έπρεπε από τη μια μεριά να πιέσουμε για να μην υπάρχουν τόσο αυστηροί στόχοι όσον αφορά την εγκατάλειψη του άνθρακα. Αλλιώς θα έπρεπε να πιέσουμε πάρα πολύ ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε υποδομές στις περιοχές εκείνες που δεν έχουν άλλες δυνατότητες να μπορούν να έχουν μια εναλλακτική πηγή προμήθειας ενέργειας. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να λυθεί περισσότερο υπόψη ότι χρειάζονται χρήματα για τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να βασίζεται όλο και λιγότερο η Ευρώπη σε χώρες οι οποίες είναι σήμερα τόσο ασταθείς ως πηγές ενέργειας. Αυτά άμα θέλουμε να φύγουμε μακριά από τον άνθρακα. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Μπόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ για τόσο μας είπατε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όπω είπατε για όλου μας. Στηρίζω απόλυτα τις προσπάθειές σας να επιταχύνουμε το έργο μας όσον αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά. Σήμερα συζητήσαμε για το ρόλο του οργανισμού ΕΝΙΣΑ και για το μέλλον του. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τον κύριο Τζακομέλη που είναι αρμόδιος και για την ασφάλεια των ε, τηλεπικοινωνιών, πώς θα βελτιωθεί το επίπεδο της ασφάλειας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ακούσει ότι ορισμένες χώρες την ε, συνεργασία την βλέπουν σαν υψηλού επίπεδου συζήτηση και θέλουν να περιοριστούν μόνο σε συζητήσεις. Εντάξει, Πρέπει και σε επίπεδο στρατηγικής να συνεργάζονται οι χώρες μέλη, όμως είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία αυτή θα γίνεται και σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Γιατί η ασφάλεια στον κυβέρνοχώρο είναι ένα τεχνικό θέμα, άρα η συνεργασία πρέπει να γίνεται και σε αυτό το επίπεδο. Τα στοιχεία κλειδί για να, εφαρμοθεί, η, να εφαρμοστεί η νέα οδηγία και να έχουμε εγγύσει για επιχειρησιακή συνεργασία θα είναι ένας πολύ σημαντικός δείχτης. Εσείς προεδρεύετε στις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο γι' αυτό, οπότε θέλω να τα λάβετε υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει μεγάλη, πολλές δυνατότητες με τις συζητήσεις αυτές που έχουμε και για την περιαγωγή και για την δετερότητα των δικτύων. Συζητάμε πολύ. Ελπίζω να μην ε, αμβληθεί το περιεχόμενο της νομοθεσίας εφεξής. Έχω δύο ερωτήσεις. Το ένα έχει να κάνει με το διοικητικό άκθος. Είναι κάπως απογοητευτικό με όλες τις φιλοδοξίες που έχετε και καλά κάνετε και τις έχετε. Δεν υπάρχει στην ατζέντα της Αλληλικής Προεδρίας η μείωση του διοικητικού άχθους. Θα έπρεπε κατά 10-15% να μειωθεί. Αν γινόταν αυτό, αυτό θα είχε αμέσως επιπτώσεις θετικές. Και το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο πάει πίσω στον τομέα αυτό, στη μείωση του διοικητικού άχθους. Καταλαβαίνω, μπορεί να μην μπορεί να είναι πρώτη σας προτεραιότητα, αλλά θα ήθελα αν μη τι άλλο να φροντίσετε να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεύτερον, κυρώσεις στη Ρωσία. Ε, σίγουρα εσείς θα δώσετε κάποια εντολή στους διαπραγματευτές σας, οπότε θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς να γίνεται η συζήτηση όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της Ουκρανικής κρίσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μπλάνκο Λόπες τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Η επαναβιομηχανοποίηση είναι πολύ σημαντικό για την απασχόληση στην ε, Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ευνοηθούν και δεν θα ευνοηθούν αν δεν υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση, πιστώσεις. Δεν δημιουργείται ευνοϊκή ατμόσφαιρα αντίθετα ακριβένει η ενέργεια όπως συμβαίνει και ελλείψη φορολογικής εναρμόνισης. Χρειάζεται λοιπόν κάτι για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες όσον αφορά την βιομηχανική της πολιτική. Προσοχή, δεν είναι καλό δείγμα οι περικοπές που είδαμε όσον αφορά τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα υποβάλω και εγώ τροπολογία από αυτού. Είναι αναγκαίο λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Γιούνκερ, να υπάρξει ένας φιλόδοξος στόχος για αναδιάρθρωση στρατηγικής σημασίας. Στο θέμα του φυσικού αερίου, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Ώστε να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο του 20% του ΕΠ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπορέλντι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τζακομέλη, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον ε, κανονισμό για τις ηλεκτρονικές κοινωνικές, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκεί είναι δυνατόν ε, να επικρατήσουν οι μεγάλοι υπάροχοι και αυτό όμως είναι εις των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, και στην κυρία Γκουίντι. Ε, κατά την άποψή σας όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική η Ιταλική Προεδρία πώς προτίθεται να παρέμβει συγκεκριμένα, πραγματικά συγκεκριμένα κύριε Υπουργέ γιατί ε, δεν νομίζω ότι ελέγχθησαν πολλά συγκεκριμένα πράγματα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι λείπει βιομηχανική Ιταλική πολιτική η οποία να μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια ευρωπαϊκή πολιτική που και αυτή είναι πάρα πολύ αδύναμη. Νομίζω ότι η Ιταλική Προεδρία ε, και η Ιταλική πολιτική ε, θα πρέπει ε, να είναι έτοιμη γιατί νομίζω ότι εδώ με μεγαλοστομίες και με λόγια δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει τη χώρα μας. Ο κύριος Τσορίνιο, επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές μας για την σαφήνεια των όσων μας είπαν πραγματικά κάνατε μια εξαιρετική διάγνωση της κατάστασης. Από όσα μας είπατε, θέλω να σας ρωτήσω, ποια θα είναι η προτεραιότητα, τι θα κάνετε κατά πρώτον, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού της Ιταλικής Προεδρίας. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Αναφερθήκατε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη για την ενεργειακή ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση. Νομίζω ότι θα είχατε πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία εάν ενισχύονταν η σύνθεση ανάμεσα στην Ιβερική Χερσόνησο και την υπόλοιπη Ήπειρο. Εδώ και χρόνια το λέμε αυτό. Αν γινόταν θα βοηθούσε πολύ. Αναφερθήκατε επίσης σε νέους στόχους για την στρατηγική της Ευρώπης για το 20. Χτες όμως συζητήσαμε για περικοπές στον προϋπολογισμό και κυρίως σε τομείς πολύ βασικούς. Και άρα δεν θα υπάρξει πιο ευνοϊκό κλίμα για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Ελπίζω λοιπόν οι προτάσεις σας να είναι εξίσου συγκεκριμένες όπως και οι ιδέες σας, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να αρκεστεί σε ωραίες ιδέες. Χρειάζεται και κάτι πιο συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέω κύριος Μαρτά. Άκουσα την Υπουργό, την κυρία Γκουίντι, με πολύ προσοχή και πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι θέλετε να προχωρήσει η Ευρώπη σε επαναβιομηχανοποίηση είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει πολύ και εμένα όλους ιδιαίτερους. Αλλά για να πετύχουμε την ε, επαναβιομηχανοποίηση, μας δούμε τι μπορεί να κάνει ο ανταγωνισμός, ο οποίος μερικές φορές παίζει το ρόλο Ταλιμπάν εντό αγωγικών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είχαμε πιο πολιτική άποψη και να είμαστε πιο ελαστικοί ώστε να αναστηθούν οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές, κυρίως σε βιομηχανικούς, στρατηγικούς τομείς, αντί να επιμένουμε τόσο πολύ στον ανταγωνισμό, ο οποίος έχει μερικές φορές καταστροφικές συνέπειες. Η Airbus, δεν θα είχε καταφέρει ότι έχει καταφέρει μέχρι τώρα, αν δεν είχαμε δράσει το παρελθόν όπως δράσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαρτά και συγγνώμη που δεν πρόφερα καλά το όνομά σας την πρώτη φορά. Ο κύριος Σκάλι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας, λέει ο κύριος Σκέλη. Κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας πριν από ένα χρόνο είχα ασχοληθεί και εγώ με τα θέματα αυτά. Δύο ερωτήσεις έχω για την ευρυζωνικότητα. Αυτό είναι ένα οικονομικό θέμα. Τι θα γίνει λοιπόν κατά την επόμενη θητεία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούν να εμπορεύονται περισσότερο online. Ευχαριστώ για την οργάνωση της διάσκεψης ε, σχετικά με τα θέματα αυτά, αλλά θα ήθελα αν μπορείτε τώρα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τα δύο αυτά θέματα. Ευχαριστούμε. Τελευταίος, η κυρία Καϊλή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ. Συγχαρητήρια για μια επιτυχημένη ως τώρα Ιταλική Προεδρία. Οι ανησυχίε όλων μα τελικά είναι κοινέ από ό,τι φαίνεται. Ήθελα απλώ να συμπληρώσω μια, ακόμα διάσταση στο θέμα τη ασφάλεια στην ενέργεια Καθώ το επόμενο τρίμηνο μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα έλλειψη και αποκλεισμού ενεργειακού από τις γειτονικές χώρες. Ε, καθώς ε, οι χώρες του Νότου έχουν υποστεί και ε, ένα, ένα σαμποτάζ, αν θέλετε να το πω, στην, στις εξαγωγές προϊόντων, αν αυτό συμβεί σε θέματα ενέργειας. Όχι απλά πώ θα τα απεξέλθουμε ω προ τι ποσότητε, καθώ υπάρχει και μια πρόταση για υγροποίηση, για υγροποιημένο φυσικό αέριο, που και στην Ελλάδα αλλά και η Ιταλία έχει αρχίσει να επενδύει σε χώρους αποθήκευσής του. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το κόστος ε, θα είναι τέτοιο που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάθε χώρα όταν έχουμε διέλθει και έχουμε εξαντληθεί σε μια πολύ μεγάλη και παρατεταμένη οικονομική κρίση. Οπότε το κομμάτι που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι αν υπάρχει και ένα πλάνο ε, για το πώς μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι που μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Και το δεύτερο κομμάτι ως προς την ε, ψηφιακή τεχνολογία ήθελα να ρωτήσω, καθώς σήμερα πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια ήταν η διαρροή προσωπικών δεδομένων και μάλιστα δεδομένων και φωτογραφιών τα οποία είχαν σβηστεί και ε, έχοντας ανέβει στο iCloud που λέγαμε ε, μπόρεσαν να υποκλαπούν και να δημοσιοποιηθούν. Μια, μια πολιτική προστασίας από την Ευρώπη, διαφορετική, χωρίς να έχει σχέση με τις εταιρείε, αλλά να υπάρχουν είτε κυρώσεις είτε μια ε, πιο σημαντική ε, ασπίδα ασφαλείας και πρόληψη για τέτοιες περιπτώσεις, καθώς να θυμίσω ότι και το, το Google έχει βγάλει ένα application στο οποίο μπορεί να παρακολουθεί κανείς ε, την καθημερινή του διαδρομή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλα αυτά τα δεδομένα, τα data μπορεί ανα πάσα στιγμή να υποκλαπούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Madame. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πιο γρήγορα από πριν, για να μην σας πάρω πάρα πολύ χρόνο. Μπονάνο, αν κατάλαβα καλά, μιλούσατε για θέματα κατά βάση Ιταλικής ε, θέσεις. Για την Νάπολη εγώ δεν θα σας απαντήσω, διότι ο συσχετισμός που κάνετε με την Νάπολη είναι καθαρά αξιολογικός και δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Για τις κυρώσεις προς την Ρωσία, το θέμα το έθιξε και ο κύριος Τέλιτσκα. Προφανώς δεν ανήκει στην δική μου αρμοδιότητα. Είναι προφανές ότι οι κυρώσεις στην κατάσταση αυτή όλοι ευχόμαστε να υπάρξει λύση. Η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε είναι να προσπαθήσουμε να υπάρξει σύγκληση θέσεων το συντομότερο δυνατό ευχόμαστε. Η Ευρώπη είναι μια αξιολόγηση που θα κάνουμε και θα παρακολουθήσουμε. Η Ευρώπη θα έχει προφανώς συνέπειες και οικονομικού χαρακτήρα. Θα υπάρχουν συνέπειες για την Ευρώπη και οικονομικού χαρακτήρα. Οι επιπτώσεις ελπίζουμε βεβαίως όλοι να μην υπάρχουν στα θέματα της ασφάλειας τουλάχιστον. Πρόκειται λοιπόν για μία μόνιμη παρακολούθηση υποστηρικτικού χαρακτήρα μιας διαδικασίας που ελπίζουμε να λυθεί θετικά. Οι επιπτώσεις αυτών των αντιμέτρων που λαμβάνει η Ρωσία θα κρυθούν από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκό σε σχέση με μια έκτακτη κατάσταση που θα πρέπει να μας οδηγήσει όλους ε, στο να το αντιμετωπίσουμε το δυνατό. Άλλα θέματα που προσπαθώ να κλείσω γρήγορα. Βλέπω ότι παρεμβάσεις ε, Γκίμπιτς, Κάρλς, ε, Φέντελε, ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Ενεργειακή ασφάλεια, διασυνδέσεις, ανανεώνυμα από, από ανθρακοποίηση, μείωση της χρήσης του άνθρακα. Εμείς και ως Ιταλία και ως ε, Προεδρία υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε βεβαίως να δουλεύουμε τόσο ώστε να προχωρήσουμε προς την μείωση της εξάρτησης από τον άνθρακα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τους υδρογονάνθρακες και τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι εις βάρος των, ε, της αποτελεσματικότητας ενέργειας και τα δύο και οι ανανεώσιμες και η απόδοση έχουν τελικό αντικείμενο τη μείωση της εξάρτησης από τον άνθρακα. Προφανώς τα κράτη και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή. Στο βραχυπρόθεσμα βέβαια πιστεύω ότι το θέμα που τέθηκε από τον κύριο Μπλάνκο Λόπες για την, τις διασυνδέσεις, τις επενδύσεις και την ενίσχυση των υφιστάμενων διασυνδέσεων με χρηματοδότηση από τα λεγόμενα έργα ευρωπαϊκού στρατηγικού χαρακτήρα. Είναι στρατηγική μέσο πρόθεσμη σε κάποιες περιπτώσεις. Βράχοι πρόθεσμα θα ενισχυθούν οι εναλλακτικές πηγές για την, τα ανανεώσιμα και την αποτελεσματικότητα στην ενεργεία θα συνοδευτούν από ορισμένε ε, ε, περιφερειακού χαρακτήρα δράσεις των ΤΑΡ, για τον ΤΑΠΕ παράδειγμα που θα έχει επιπτώσει στην Βαλκανική Χεσόνησο, θα γίνουν κατόπιν στρατηγικά για την ενίσχυση των διασυνδέσεων, ούτω ώστε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα και μια δέσμη άλλων πηγών. Υγροποιημένο αέριο, για παράδειγμα. ενισχύοντα κάποιε διασυνδέσει, για παράδειγμα, που σήμερα λείπουν. Π.χ. μεταξύ Ισπανία και υπόλοιπη Ευρώπη. Σε μια οπτική ευρωπαϊκή, συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική. Και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που έλεγα στην αρχή είναι το εξής. Ως Ιταλία πιστεύουμε πολύ στο Industrial Compact που ξεκινήσαμε και σε ιταλικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να έχει η Ευρώπη μια βιομηχανική στρατηγική που θα δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο. Πιστεύω αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Το mainstreaming της ανταγωνιστικότητας βιομηχανίας είναι καθοριστικό για να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ε, βιομηχανική βάση που θα είναι ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική. Πιστεύω λοιπόν ότι σε ε, επίπεδο προεδρίας είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουμε τις ε, ενδείξεις που έδωσε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου να υπάρξει ένας ε, οδικός χάρτης, ένα roadmap που θα συνδέεται στην ανάγκη ενός mainstreaming της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης και των βασικών θεμάτων και σημείων στα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση ακριβώς για να ξαναδώσουμε ε, όθηση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ικανότητες, τις ίδιες ικανότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι που πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη μας να δημιουργήσουμε δηλαδή Ευρωπαίους πρωταγωνιστές, Ευρωπαίους πρωταθλητές σε κάποιους τομείς. Το έλεγα το πρωί σε μια συνάντηση με τους Ιταλούς Ευρωβουλευτές. Κάποια από τα θέματα της αποβιομηχανοποίησης που βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οφείλονται εν μέρη και στον ανταγωνισμό που προέρχεται από έξω από την Ευρώπη. Πρόκειται για ανταγωνισμό που συχνά, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον, δεν είναι πολύ fair, πολύ θεμητή, θεμητές μορφές ανταγωνισμού. Γιατί έρχονται από τρίτες χώρες και σε κάποιους στρατηγικούς τομείς, βασικούς και για τις χώρες αλλά και για την Ευρώπη, Φερρυπίνο Χάλιβας, τα τελευταία χρόνια υπέστησαν τελείως αθέμητη, αθέμητο ανταγωνισμό από εξοκοινωτικούς ανταγωνιστές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Πρόσβαση λοιπόν σε χρηματοδοτικούς πόρους, υποστήριξη όλων των παραγόντων που ενισχύουμε, ευχόμενοι αυτό το roadmap να αποτελέσουν την πηξίδα των δράσεών μας. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα επιχειρήματα. Thank you very much, Madam. Madam Minister, and I would like to ask for... Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Τώρα ο Υφυπουργός να απαντήσει στις τελευταίες ερωτήσεις, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπατε σχετικά με την οδηγία ενής. Για μας ε, είναι μια προτεραιότητα της ε, Προεδρίας μας. Συνεργασία να υπάρχει όχι μόνο σε στρατηγικό αλλά και σε επιχειρησιακό τεχνικό επίπεδο. Συμφωνώ επ' αυτού. Προφανώς ε, δεν ήρθα εδώ για να εκφράσω μόνο τη δική μου άποψη. Ε, έχω υπόψη μου τη δουλειά που πρέπει να γίνει έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να επιδιώξουμε τους στόχους μας. Βεβαίως και τα ε, συστήματα προστασίας διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος. Εμείς η Προεδρία έχουμε προτείνει ένα νέο κείμενο στην ομάδα εργασίας και στόχος είναι να υπάρξει ένας κοινό μηχανισμός για να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνοαπειλές. Οι απειλές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην αξία της στρατηγικής συνεργασίας. Βεβαίως και είναι σημαντικό να φτάσουμε εκεί, αλλά αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο είναι να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το επίπεδο των δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσονται. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο είναι σημαντικό να ε, σφυριλατηθεί μια προοδευτική σχέση συνεργασίας. Η οδηγία ΝΙΣ ε, ελπίζουμε ότι θα ε, τελεσφορήσει κατά τη διάρκεια της δικής μας της ε, Προεδρίας. Τώρα, όσον αφορά στην περιαγωγή, πρέπει να σας πω, δεν έχουμε καμία πρόθεση να δεχτούμε αυτή την άποψη που προέκυψε τόσο από την έκθεση της κυρίας Κρούζ όσο και από την ε, εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντική η δουλειά της Προεδρίας με την έννοια ότι η δουλειά αυτή βοηθάει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να διεκδικήσουν όλα τον ίδιο στόχο. Και το μήνυμα που ε, θα πρέπει να περνάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα σαφές μήνυμα για μια κοινή πολιτική, για μια ε, ουσιαστική ψηφιακή πολιτική. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν να ε, νοθεύσουμε την πολιτική, αλλά σε κάποια κράτη υπάρχει ένα σχεδόν αυτόματος μηχανισμός του συστήματος ε, περιαγωγής. Και αυτές οι κυβερνήσεις ε, αντιμετωπίζουν με ανησυχία ε, τις εξελίξεις γιατί για αυτές είναι μια εικονική διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ούτε ε, πρέπει να μπλοκαριστούμε από όλα αυτά, αλλά ούτε και να αγνοούμε τις εξελίξεις. Ε, να φτιάξουμε όμως τους απαραίτητους μηχανισμούς, γιατί ε, πράγματι είναι σημαντικό να μην υπάρχει περιαγωγή, να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και όλα αυτά πρέπει να γίνουν από κοινού και κοινά τα προβλήματα, από κοινού πρέπει να ζητηθούν και λύσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Μπορέλη. Ε, το θέμα των ε, δικτύων είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Όταν μιλάμε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και όλες αυτές οι ευκαιρίες που ε, προσφέρει το διαδίκτυο. Έχουμε κατά νου ένα διαδίκτυο που προσφέρει ευκαιρίες που δεν περιορίζει τις ε, θετικές ε, επιπτώσεις και τα θετικά στοιχεία μόνο σε όσους έχουν οικονομική ευμάρεια. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή στην Αμερική μιλάνε σαν να υπάρχει ε, κάποιο είδος συγκερασμού εξελίξεων και επιτροπών. Τα ήθελα βέβαια να μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Τζορίνιο. Θα μπορούσα να του πω τελικά με τι πρέπει να ξεκινήσουμε ή ε, θα μπορούσαμε να μπορώ να σας πω ε, το τι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος. Η εννέα ψηφιακή αγορά, ε, το θέμα της ε, governance, ε, η ουδετερότητα του δικτύου. Ίσως θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα-δύο πράγματα και τα άλλα να τα αναβάλουμε. Αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε εμά, αλλά οφείλεται κυρίως στην ευρωπαϊκή διάσταση. Επ' αυτού νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να ε, ενώσει τους τις προσπάθειες λόγω της ιστορίας της και της παράδοσης ε, να δούμε τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό το σενάριο και τις ε, δυνατότητες επενδύσεων. Αυτά όλα μπορούν να παίξουν σημαντικό όλο σε διεθνές επίπεδο και αυτό θα βοηθήσει τα μάλα την ψηφιακή επανάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι οι σωστές ε, απαντήσεις. Τα κράτη-μέλη, εάν το Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις, αν όλοι μαζί αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, νομίζω ότι τη φιλοδοξία που σας ανέφερα μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Κύριε Κέλλη, το ηλεκτρονικό εμπόριο αυτό δεν είναι στις άμεσες αρμοδιότητές μας, αλλά νομίζω ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ίσως ε, μπορούμε να σκεφτούμε το τι ακριβώς ε, πρέπει να εφαρμόσουμε. Ένα θέμα επί το οποίο ε, πρέπει να εμβαθύνουμε. Οι στόχοι για την Internet Governance αυτούς τους ανέφερα. Η ιδέα ότι το άτυπο συμβούλιο των Ευρωπαίων κρατών ε, θα πρέπει να συμμερίζεται αυτή την ε, προσέγγιση που υπάρχει με βάση την ε, ICAN και με βάση κάποιες αρχές την ελευθερία έκφραση, την ελευθερία δημιουργίας, το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας Αυτά πρέπει να είναι τα σημεία επί με βάση τα οποία μπορεί κανείς να επιδιώξει ένα νέο μοντέλο governance. Να δείξουμε στην Ευρώπη ότι υπάρχει μία ενιαία φωνή, κυρίως στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν είναι ανησυχητικά και απευθύνομαι στην κυρία Καηλή όχι μόνο όσον αφορά τη διαρροή των ατομικών δεδομένων, αλλά κυρίως για το τι αποκαλύπτουν όλα αυτά. Σήμερα ε, νομίζω βλέπουμε όλοι ότι πολύ εύκολα έρεται και καταργείται η ιδιωτική σφαίρα. Ακόμα το διαδίκτυο δεν είναι σε θέση να προστατεύσει πλήρως όλους τους πολίτες την ιδιωτική σφαίρα των πολιτών. Δεν είναι ότι για μας η δική μας αρνητοδιότητα δεν είναι να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες κυρώσεις, αλλά να επιμείνουμε στο ότι η προστασία της ποιητικής σφαίρας είναι αναφέρατο και αναλύωτο δικαίωμα και αν θέλετε αυτό είναι και ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Κύριε Υφυπουργέ. Θα το έχετε καταλάβει από τις παρεμβάσεις μας ότι έχετε στήριξη στις προτεραιότητές σας και σε ό,τι κάνετε. Τους επόμενους τέσσερις μήνες μόνο έχουν μείνει και πρέπει να αφαιρέσουμε και τις, τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, δηλαδή μισή μήνες ουσιαστικά σας μένουν. Πάντως σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Οι προτεραιότητές σας είναι πολύ σημαντικές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ακούσαμε και η Επιτροπή μας Ήτρε προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την Ιταλική Προεδρία. Οπότε περιμένουμε να έχουμε ξανά συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστούμε λοιπόν για το χρόνο που μας διαθέσατε. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ και πάλι. Και σταματήστε τα πηγαδάκια. Παρακαλώ. Εσείς εκεί. Είμαι Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτησή μας με την κυρία Στεφανία Τζανίνη, που είναι Ιταλίδα Υπουργό Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας. Εκπροσωπεί εδώ την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Η κυρία Στεφανία Τζανίνη αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Πίζα και της Πάντουα και έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Έχει μεγάλη λοιπόν ακαδημαϊκή πείρα. Ήτανε μάλιστα και πρίτανης στην Περούτζια. Ασχολήθηκε με την εκπαίδευση τον πολιτισμό και ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης για την έρευνα, την ηθική και την βιοηθική του Ιταλικού Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου. Ήταν και εκπρόσωπος της διάσκεψης των Πριτάνεων των Ιταλικών Πανεπιστημίων. Πολλά έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία και εξελέγει και γερουσιαστής το 2013. Ήταν επικεφαλής της Επιτροπής του, της Γερουσίας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Είναι εδώ πρόσωπος της Ιταλικής Προεδρίας για ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι η έρευνα και η καινοτομία. Στο χαρτοφυλάκιό της είναι κοινέ τεχνολογίες και η σύνδεση της βιομηχανικής με τις ακαδημαϊκές κοινότητες. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καλή σας, πολύ ευγενική παρουσίασή σας. Θα μιλήσω Ιταλικά. Λόγω της θέσης μου και του ρόλου μου. Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε. Κύριοι και κυρίες συναδελφοί, είναι τιμή και προνόμιο για μένα να είμαι εδώ παρόν στην Επιτροπή σας που ευχαριστώ για τη διατρισμόσυντα που δείξατε, ούτως ώστε να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες του Ιταλικού εξαμήνου στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και του διαστήματος. Έχω επίγνωση, έχουμε επίγνωση της ε, ευθύνης που η Ιταλία ως ε, έχουσε την προεδρία της Ένωσης έχει. Ε, με δύο σημαντικές περιπτώσεις, πιο σημαντικά. Πρώτον, την νέα, τη σύμπτωση τις προεδρίας μας με το νέο επταετές πλαίσιο και το Horizon 2020 στη χώρα μας, στην Ιταλία, ανατέθηκε ευθύνη, άρα και η ευκαιρία να δώσουμε στρατηγικές γραμμές για να γίνουμε υπεύθυνοι της στρατηγικής της Ένωσης σε κρίσιμους τομείς, αυτούς που είναι βασικοί για το μέλλον της Υπήρου μας, της Ευρώπης που επιτρέπει ανάπτυξη και πρόοδο. Η δεύτερη στιγμή είναι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το πέρασμα μεταξύ της παλιάς και της νέας επιτροπής που ξεκινά τον Νοέμβριο του παλαιού και του νέου κοινοβουλίου που εκπροσωπείτε εσείς εδώ. Στο πλαίσιο αυτό, ευθύνη μας είναι να δουλέψουμε με αποφασιστικότητα και δέσμευση σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο αλλά και τις αρμόδιες ε, επιτοπές. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όχι μόνο δική μου, αλλά ολόκληρη της Ιταλικής Προεδρίας, ότι το υφιστάμενο πλαίσιο κρίσης ε, δεν, είναι, δεν εκπροσωπεί μια συγκυριακή ή μεταβατική φάση, αλλά και αποτελεί μια περίοδο παραδειγματικής αλλαγής που πρέπει να καταγράψουμε και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε πολιτισμικό επίπεδο και δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι οι επενδύσεις σημαντικές στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε καλύτερα αυτή την αλλαγή παραδείγματος δίνοντας τις σωστές απαντήσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε πολύ σημαντικές τις προτάσεις για ένα πρόγραμμα επενδύσεων που πρότεινε ο κύριος Γιούνκερ. Είναι δύο τομείς, έρευνα και ανάπτυξη, που έχουν στρατηγικό ρόλο. Έρευνα σημαίνει επένδυση με σαφείς καθοριτήριες γραμμές, ούτως ώστε να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, με στέρεες υποδομές που θα είναι hub για επενδύσεις στην κατάρτιση. Το λέμε συχνά, αλλά δεν είναι εύκολο να το ελοποιήσουμε. Σημαίνει να κάνουμε την ευρωπαϊκή κοινωνία καλύτερα εκπαιδευμένη με ικανότητες που θα κάνουν τους νέους μας να αποκτήσουν την απαραίτητη επαγγελματικότητα για τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους. Το βασικό λοιπόν στοιχείο της προεδρίας μας συνδέεται με αυτή την συνολική προσέγγιση που έχουμε. Επαναλαμβάνω ξέρετε ίσως, ανάπτυξη και απασχόληση πρώτον, χώρος ελευθερίας ασφάλειας για πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων πολίτη δεύτερον και ένας ισχυρότερος ρόλος, στρατηγικός, περισσότερο στρατηγικός ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο. Στην διαμόρφωση των προτεραιοτήτων αυτών σε έναν τομέα έρευνας και καινοτομίας μπορώ να σα πω ότι προφανώ εμπνευσήκαμε και ενσωματωθήκαμε σε αυτό το τριώνυμο των προτεραιοτήτων. Ξεκινώ από ένα σημαντικό θέμα, τις υποδομές έρευνας. Στις 22 Ιουλίου άλλωστε για το θέμα αυτό είχαμε μια άτυπη συνάντηση των Υπουργών Έρευνας, αυτό είναι και παράδοση. Και παράδοση. Στη συνάντηση αυτή την προσοχή μας, την επικεντρώσαμε σε, τρεις, σε τρία βασικά θέματα. Στρατηγικός προγραμματισμός τους, ο ρόλος δηλαδή του European Strategic Forum, που είναι το κέντρο βάρους του προγραμματισμού και των ενδείξεων των αρχών στον τομέα των ε, υποδομών αυτών, την βέλτιστη χρήση optimization των εθνικών πόρων και των ευρωπαϊκών πόρων για να βρούμε μηχανισμούς που είναι πραγματικά ικανοί να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν την αριστεία και το ταλέντο. Τέλος, την βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα για να έχουμε μία ανοιχτή προσέγγιση των υποδομών έρευνας προς την κοινωνία και τον κόσμο, ανοίγοντάς τον στον παραγωγικό κλάδο. Τους επόμενους τέσσερις μήνες έχουμε δύο σημαντικά συμβούλια υπουργών έρευνα κατά ε, την προεδρία μα 26 Σεπτεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου και θα ασχοληθούμε κατά βάση και με τι θεματικέ αυτέ. Έχουμε την πρόθεση να προτείνουμε μια πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου εν ώψη των συμπερασμάτων που μπορούν να προκύψουν από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας ως πηγές ανάπτυξης ποσοτικά και ε, αύξηση μεγέθυνσης ποσοτικά και ανάπτυξης ποιοτικά της Ένωσης. Βάση και μιας ε, ανακοίνωσης επιτροπής για το θέμα αυτό. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να είναι βασικά θεμελιώδη στοιχεία, ούτω ώστε τη δραστηριότητα μα για να μπορέσουν τα συστήματα παραγωγή να περάσουν προ ένα πιο έξυπνο smart specialization το λέμε, ένα πιο έξυπνο μοντέλο ανάπτυξης που θα είναι και βιώσιμο και συμπεριληπτικό. Πρόκειται για τρεις λέξεις που πρέπει να υπογραμμίζουμε. Έξυπνο, βιώσιμο, συμπεριληπτικό. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την αναθεώρηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020. Ε, η Προεδρία εκεί θα δώσει μεγάλη σημασία. Οι βασικές ε, πτυχές που θέλουμε να τονίσουμε είναι η αιτιώδη σχέση που πρέπει πάντα να υπογραμμίζουμε μεταξύ έρευνας και καινοτομίας, αναγκαίο για να βελτιώσουμε το οικοσύστημα της καινοτομίας, ο συντονισμός μεταξύ εθνικών ερευνητικών συστημάτων και ευρωπαϊκών ερευνητικών συστημάτων, σύνδεση των εθνικών προγραμμάτων έρευνα και μεγάλων προκλήσεων όπως αυτές που περιλαμβάνει το Horizon 2020, ιδίως ένα σημαντικό καθοριστικό θέμα που είναι η πραγματική δυνατότητα να υπάρξει μια κινητικότητα ερευνητών και νέων ε, ε, επιστημόνων. Και τέλος η χρησιμοποίηση των επενδύσεων έρευνας και κοινοτομίας με καλύτερο τρόπο μέσω της σύνδεσης δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας. Αυτό το μοντέλο δημόσιο-ιδιωτικό που πρέπει να επανεξεταστεί και να χρησιμοποιηθεί αυτές. Οι Joint Technology Initiatives, για παράδειγμα, που ξεκίνησαν εδώ στις 9 Ιουλίου, μου... και είχα την τιμή να είμαι και παρούσα. Είναι ένας από τους άξονες που μπορεί να πάρει ο δρόμος αυτός. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε μια παγιωμένη πολιτική συνένεση, ούτω ώστε όλα αυτά να υλοποιηθούν στην ευρωπαϊκή πολιτική έρευνα των επόμενων ετών. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε την γεωπολιτική παράμετρο του θέματος. Μια άλλη προτεραιότητα της Ιταλικής ε, Προεδρίας, ε, η διαμόρφωση δηλαδή μιας μεγάλης στρατηγικής πρωτοβουλίας, ε, εταιρικής σχέσης για την έρευνα και καινοτομία με τις χώρες της Μεσογείου. Ακολουθήσαμε εδώ τα εξαιρετικά αποτελέσματα που μας παρέδωσε η ελληνική προεδρία. Θέλουμε να λανσάρουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area, το πρίμα ε, με το ακρόνιμο, που έχει στόχο να επεξεργαστεί δύο βασικούς ε, τομείς, το νερό και τα τρόφιμα στο γενικότερο κλάδο της επιστημιστικής ασφάλειας για να δημιουργηθεί ένα μοντέλο στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των ερευνητικών Ινστιτούτων ε, της Μεσογείου. Στο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια σχετική συζήτηση προετοιμάζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου για το ζήτημα. Με στόχο να έχουμε ένα νέο κοινό πρόγραμμα βάσει το άρθρο 185 τη συνθήκη για το θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου εδώ κυρίες και κύριοι, να ζητήσω την υποστήριξή σας, γιατί θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεδομένου, δεδομένης της στρατηγικής αξίας και της σημαντικής προοπτικής που αυτό το πρόγραμμα θα έχει, καθώς και των επιπτώσεών του γεωπολιτικά, για να δημιουργήσουμε μια ειδική υποδομή έρευνα στην περιοχή αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης έχει καθοριστικό ρόλο και εδώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις στην διαμόρφωση αυτής της λεγόμενης science diplomacy. Για τη Μεσόγειο πάντα θέλουμε να υπογραμμίσουμε και να αναδείξουμε το θέμα της ανάπτυξης των ενάλιων δραστηριοτήτων, της λεγόμενης μπλε ανάπτυξης ε, που αφορά όχι μόνο τις μεσογειακές χώρες αλλά και άλλες και που θα επιτρέψει να υπάρξει μεγαλύτερη ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία στην περιοχή αυτή. Τρεις διασκέψεις θα γίνουν σχετικά στη Ρώμη ε, τον Σεπτέμβριο, στο Τωρίνο για την βιοοικονομία και τον Νοέμβριο στην Νάπολη για την εξέλιξη της ενάλλειας οικονομίας. Τρίτη προτεραιότητα στον τομέα αυτό της έρευνας είναι η ολοένα και περισσότερο αναγκαία σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Υπάρχει μια κοινωνία που χρειάζεται την επιστήμη, που είναι έτοιμη να τη δεχθεί. Ταυτόχρονα ο επιστημονικός κόσμος είναι έτοιμος να ανοιχτεί, σπάζοντας και κάποια εμπόδια του παρελθόντος, προς την κοινωνία. Για το σκοπό αυτό προγραμματίσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για θέματα κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θέματα που ξεκινούν από μια σαφή ένδειξη της πολιτικής της Επιτροπής. Τα θέματα που θέλω να τονίσω αφορούν τις έξυπνες κοινότητες, την ανάδειξη του της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ε, κλιμακότητα της κοινωνικής κοινοτομίας και επιστημονικά και, χρηματοδο... και τεχνολογικά και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής κοινοτομίας, ένα καινούριο θέμα σημαντικό που πρέπει να εντάξουμε στην θεματική. Για το λόγο αυτό θα γίνει μια ειδική διάσκεψη στη Ρώμη μεταξύ 19 και 21 Νοεμβρίου για το μέλλον της επιστήμης με και για την κοινωνία. Κάτι που θα επιτρέψει και στο τέλος του εξαμήνου μας να έχουμε μια έτοιμη συλλογιστική για το θέμα αυτό. Και όσοι θέλετε από εσά, με χαρά να σας δούμε και στην εκδήλωση αυτή. Αυτά, συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν μόνο αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο έρευνας βάσει των οδηγιών που έχουμε, από τις οποίες ξεκινήσει, που δείχνουν την βασική κατεύθυνση της στρατηγικής Ευρώπης το 2020. Αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος είναι βασικό εργαλείο και για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, των νέων ερευνητών για παράδειγμα, όσο και διότι η γνώση και οι ιδέες πρέπει να μπορούν να γίνουν κοινή κληρονομιά και όχι μόνο ιδέες. Για το στόχο αυτό, υπενθυμίζω, συνθετικά κάποιες βασικές λέξεις που σίγουρα είναι γνωστές σε όλους και που θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία της δουλειάς. Κινητικότητα. Κινητικότητα ερευνητών, πρόσβληση με βάση κοινού ανοιχτούς και διάφανους κανόνες και διασυνοριακή συνεργασία που μπορεί να γίνει μια ενάρετη ευκαιρία σύνδεσης μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και όταν μορφώνουμε το εθνικό πρόγραμμα έρευνας στις χώρες μας. Ένα σημαντικό κείμενο που ετοίμασε το κοινοβούλιο σας πέρυσι το 2013 που στο οποίο δούλεψαν οι Ιταλοί ευρωβουλευτές κυρία Σαρτόρη και Μπεριλγορή και που έχει τον τίτλο «Μάστρεχ της έρευνας» συμβάλλουν ιδιαίτερα στις εργασίες μας αυτό. Και γι' αυτό 18-19 Νοεμβρίου θα ετοιμάσουμε στο Τρέντο μία εκδήλωση ακριβώς για την πρόθεση της αριστείας και την κινητικότητα και στην πρόσληψη. Αυτή λοιπόν η ιδέα ότι οι stakeholders είναι καθοριστικά στοιχεία της ε, κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η ιδέα με άλλες ε, που αφορούν ε, περισσότερο ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες. Αυτά θα μπορούσαν να είναι οι πρωταγωνιστές σε μια, μιας πραγματικά ελεύθερης αγοράς. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να προάγουμε. Βεβαίως... Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός χώρος έρευνας ε, και κινδυνεύουμε όλα αυτά να γίνουν πολύ αφηρημένα αν δεν έχουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε. Το πρώτο είναι το ότι τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να ε, ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις ε, που είναι γύρανση του πληθυσμού, το θέμα της ε, μετανάστευσης, η κινητικότητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει κάποια σχέση σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια των κρατών μελών και αυτήν της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, οι προκλήσεις αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν. Έχουμε δυστυχώς δραματικά παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Προεδρία ε, θα μπορέσει να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με βάση όλα αυτά που σας ανέφερα ε, στο Συμβούλιο της 21ης Σεπτεμβρίου με στόχο να εγκριθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα στο Συμβούλιο πλέον του Δεκεμβρίου. Έχω νομίζω άλλα δύο-τρία λεπτά στη διάθεσή μου για να σας ε, μιλήσω και να αναφερθώ σε ένα θέμα ε, που το αναφέρω στο τελευταίο αλλά σίγουρα δεν είναι έσχατο. Είναι το θέμα της διαστημικής έρευνας. Το διάστημα και αυτό είναι ένας από τους ε, τομείς ε, όπου πραγματικά διακυβεύεται η πρόοδος της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο. Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική ε, τόσο κάτω από το πρίσμα των κοινών, κοινοτικών πολιτικών όσο και των βεβαιωμένων εθνικών πολιτικών είναι μια καθοριστική, πολύ σημαντική πολιτική. Είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Ε, Δεν έχουμε προχωρήσει δυστυχώς στον τομέα αυτό όσο θα επιθυμούσαμε. Το θέμα λοιπόν του διαστήματος έχει άμεση σχέση και με θέματα χρηματοδότησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ε, η Ευρωπαϊκή, η Ιταλική με Προεδρία, εμείς θα λάβουμε υπόψη μας κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, σύντομα, πρώτον είναι η ενίσχυση των ε, στρατηγικών των διαστημικών ε, πολιτικών, αξιολογώντας επενδύσεις του παρελθόντος, αλλά και βελτιστοποίηση των επενδύσεων που θα γίνουν κατά επόμενα 7 έτη. Υπάρχουν όμως και άλλα πολύ συγκεκριμένα θέματα και θέλω να σας υπενθυμίσω για τα επόμενα 7 έτη έχουν προβλεφθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Γαλιλαίο Έγνος, για το Κοπέρνικους και για την έρευνα στο διάστημα. Πρόκειται λοιπόν για μια ε, πρωτοφανή αύξηση η οποία είναι ερευνητικής φύσεως αλλά και οικονομικής και πολιτικής και αφορά το, όλο το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Η δική μας η πρωτοβουλία είναι το να προωθήσουμε την οδηγία για τον εντοπισμό, ε, την, τον εντοπισμό των ε, δεδομένων, των γεωσκοπικών δεδομένων και ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδώσουμε στην ε, στρατηγική σημασία που μπορεί να έχει η ανεξαρτησία στη συλλογή και εντοπισμό αυτών των δεδομένων και στη χρήση τους για στόχους που δεν είναι μόνο αμυντικοί, στρατιωτικοί, αλλά στόχοι που μπορούν να εφαρμοστούν και στην κοινωνία. Ε, το διοικό αυτό μοντέλο το έχουμε κατά νου. Αυτό προέκυψε από το πρόγραμμα Cosmos SkyMed. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν ως στόχο να προετοιμάσουμε μια ε, πολιτική που θα έχει στόχο το μέλλον της σχέσης ε, με την ε, ευρωπαϊκή πολιτική και την διαστημική πολιτική. Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα διάλογο από κοινού με την ΕΖΑ για να ορίσουμε ποια, ποιες θα πρέπει να είναι οι σχέσεις, οι νέες σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την, ε, τον Διαστημικό Οργανισμό. Ως Προεδρία θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα και να παίξουμε καθοριστικό ρόλο ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε με απόλυτη στράτευση. Μία άλλη πρωτοβουλία που θέλω να σας ε, αναφέρω είναι αυτή του, της 18 Σεπτεμβρίου, μία συνάντηση που θα λάβει η χώρα στη Ρώμη και θα αφορά η πρωτοβουλία αυτή το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Μιλάμε για μία σημαντική μετάβαση από την βασική έρευνα ε, σε επίπεδο διαστημικό. Τέλος, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι ένα θέμα που βέβαια αφορά περισσότερο ε, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας. Θέλω όμως να αναφερθώ εκ μέρους της Ιταλικής Προεδρίας στη δέσμευσή μας για την ε, συνεχιζόμενη εφαρμογή των προγραμμάτων Γαλιλαίος σε σύστημα, σύστημα, παγκόσμιο σύστημα ε, πλοήγησης μέσω των δορυφόρων. Θα κάνουμε αυτό που προβλέπετε και γνωρίζουμε πολύ καλά το ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για τα κίνητρα, τα αίτια τα οποία οδήγησαν ε, σε ένα δυστυχές ατύχημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, προσοχή σας και θα ήθελα με αυτά τα λόγια να ολοκληρώσω επισημένοντας ότι ελπίζω αυτά τα θέματα να είναι πολιτικά σημαντικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, κύριε Υπουργέ της Ιταλικής Προεδρίας όσον αφορά το διάστημα κλπ. Ψηφίσαμε τον ετήσιο προπολογισμό μας για την επόμενη χρονιά της τροπολογίας μας μάλλον επί του προπολογισμού αυτού και ζητήσαμε περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σημαίνει ότι τα φροντίζουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, ας ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές μας. Ο κύριος Κάριντς, εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζανίνη, για την τόσο ενδιαφέρουσες και λεπτομερείς επεξηγήσεις που μας δώσατε για τους στόχους σας. Τις τελευταίες μέρες στην Επιτροπή αυτή Συζητάμε κυρίως την ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Είδαμε λοιπόν την, στη τη στην ψηφιακή ατζέντα, την ενέργεια, μιλήσαμε πολύ για την βιομηχανία και για τη σημασία της επαναβιομηχανοποίησης της Ευρώπης προκειμένου να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Αναφερθήκαμε στην οδηγία για την ε, διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων και όπως είπε ο κύριος Μπούζεκ, σήμερα το πρωί ψηφίσαμε τον προπλησμό για το 2015, όπου διαπιστώσαμε με θλίψη ότι πολλές φορές μέλη, περισσότερες, μειώνουν τα κονδύλια που απευθύνονται σε ερευνητικά προγράμματα, κάτι το οποίο αποτελεί ακρογωνία λίθο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Η απάντηση μπορεί να μην είναι απλή. Είπατε ότι το ρίζων 2020 αποτελεί έναν νέο τρόπο σκέψης. Εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή αυτή έχουμε δουλέψει πάνω στη σχετική νομοθεσία για τρία χρόνια και ρωτάω κατά τη γνώμη σας ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα προκειμένου να πάμε στο νέο Ορίζον 2020. Είναι μόνο θέμα νοτροπίας, είναι κάτι πρακτικό, υπάρχουν πολλές αντιστάσεις. Και τι βήματα θα αναλάβει η Προεδρία σας για να ε, τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να διατηρήσουμε έτσι την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όσο μπορούμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κρυμπάρισικ τώρα εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πολύ σύντομα. Αναφερθήκατε στην ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας στις προηγμένες τεχνολογίες και είπατε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στην κατάρτιση των νέων. Ποια είναι η λύση των νέων προκειμένου από την ανεργία να ξεφύγουν και να βρουν δουλειά. Ανεργία που είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα σήμερα. Τι θα κάνετε ώστε οι νέοι αυτοί να μην μείνουν χωρίς μέλλον. Για μένα χρειάζεται εκπαίδευση, για μένα αυτή είναι η λύση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεμπάκερ εκ μέρους της Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ ενθουσιώδης ε, όσον αφορά τις διάφορες προτεραιότητες που θα έχετε τους επόμενους μήνες μπροστά σας. Θα αρχίσω και με τις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι δηλαδή σήμερα που δημοσιονομικά βρισκόμαστε σε στενότητα σε πολλές χώρες μέλη, οι επενδύσεις στην έρευνα έχουν μειωθεί σε διάφορες χώρες και δεν πλησιάζουμε το στόχο του 3% που έχουμε θέσει. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν κίνητρα ή βήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν, συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Εξάμενο για παράδειγμα ή κάτι άλλο, ώστε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο 3%. Όσον αφορά το Horizon 2020, το συζητήσαμε ήδη για τα σχετικά κονδύλια, μια από τις κύριες προτεραιότητες δεν είναι μόνο να υπάρχει υψηλή δίκευση, αλλά να είναι πιο εύκολο για τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες κυρίως, να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια αυτά. Το είπε και η κυρία Κουίν. Πώς θα γίνει αυτό όμως στο στάδιο της εφαρμογής, η χρηματοδότηση και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη, πώς θα γίνει πιο απλή και πώς θα έχουν πιο εύκολα πρόσβαση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κονδύλια, γιατί έχουμε πραγματογνωμοσύνη να μοιραστούμε μεταξύ μας για τέτοιου είδου προγράμματα. Και Τέλος, η έρευνα για την έρευνα δεν φτάνει. Πρέπει να φτάνει στην αγορά. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσει την έρευνά μας αυτή η βιομηχανία. Τι θα κάνετε λοιπόν για να φτάσουμε σε επίπεδα άλλων χωρών, μερικών εντός αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η έρευνά μας να καταλήγει στην αγορά πώς φροντίστε να υπάρχει κάποια ισορροπία για να οδηγήσουμε την έρευνά μας στο εμπόριο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σέσενικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου ε, πρότεινε μείωση του προϋπολογισμού του ορίζον 2020. Εσείς αναφερθήκατε στη βιωσιμότητα, στην ευφία, στην ανταγωνιστικότητα, ίσως για να δικαιολογήσετε τις περικοπές αυτές. Όμως, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο διαπιστώνουμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται προσφέρει 7 με 14% προσθεθέμενη αξία στην βιομηχανία. Τώρα που υποφέρει τόσο το ευρωπαϊκό ΑΕΠ και υπάρχει τόσο μεγάλη ενεργεία, έστω και μια μικρή αλλαγή θα βοηθούσε. Εννοείται ότι πρέπει να γίνονται επενδύσεις στην έρευνα. Γι' αυτό και βρίσκω ότι είναι επικίνδυνο αλλά και απαράδεκτο αυτό που προτείνει το Συμβούλιο. Και σας ρωτάω, εσείς κύριε Υπουργέ, συμφωνείτε με τη στάση αυτή παρέτησης από την καινοτομία της Υπήρου μας. Και πείτε μας ναι ή όχι, η, Ιταλική Προεδρία θα στηρίξει τις περικοπές αυτές του Συμβουλίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η FFDD, ο κύριος Ταμπουράνο. Κυρία Τζανίνη, όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της παιδείας, της ε, τρίτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας έχουν μια ιδιομορφία. Ε, το θέμα είναι ότι θα πρέπει κανείς να συμβάλλει ε, στην ευημερία της χώρας του. Αυτή είναι η βάση για να υπάρχει πλήρης δημοκρατία. Να γνωρίζει ε, κανείς ε, το πώς πρέπει να εκπαιδεύσει τους νέους. Εμείς προερχόμαστε από μια χώρα όπου στην Ιταλία οι γονείς είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν το χαρτί τουαλέτας για τα σχολεία. Και εσείς λοιπόν λέτε ότι τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται από την Τρόικα, δηλαδή από την ΕΚΤΑ, από την Επιτροπή και από το Διεθνές Δομιστικό Ταμείο, αυτή η Τρόικα που υπάρχει στις χώρες που γνωρίζουμε μεταξύ των άλλων στην Ελλάδα θα πρέπει να επέμβει, πιστεύετε θα πρέπει να επέμβει η Τρόικα και στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε. Έχω άλλες τρεις παρεμβάσεις. Ο κύριος Τελίτσκα πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τη λεπτομερή σας παρουσίαση και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχω μία παρατήρηση σε σχέση με κάτι που αναφέρατε. Την αναθεώρηση της στρατηγικής 2020. Θα ήθελα να γνωρίζω εσείς ως Προεδρία, εσείς προσωπικά πώς βλέπετε μια τέτοια αναθεώρηση. Για να το πω μα, το μεγαλύτερο έλλειμμα της στρατηγικής 2020 είναι ότι πρόκειται για έναν κατάλογο επιθυμιών για να ικανοποιηθούν όλοι. Δηλαδή ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πάντα, χωρίς να βάζει προτεραιότητες. Δεν θα σας πω ποια είναι η δικιά μου άποψη, αλλά θέλω να ξέρω ποια είναι η δικιά σας και ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της εμπορίας. Η δυσκολία που έχω με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ταπάνες της στην καινοτομία είναι ότι δεν υπάρχει μέτρηση. Λίγο πριν από λίγο χρόνια που είχα και περισσότερα μαλλιά από αυτά που έχω τώρα, αξιολογούσαμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε τότε είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαπανούμε πλήρως τα χρήματα και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με δωροδοκίες κλπ. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε μέτρηση και νομίζω ότι ούτε τώρα γίνεται μέτρηση για να ξέρουμε πόσο βοηθούν στην καινοτομία τα διάφορα προγράμματα. Θα μπορούσαμε να εισακάγουμε λοιπόν και αυτό το στοιχείο της μέτρησης αν επενδύοντας χρήματα έχουμε πετύχει το στόχο μας ή όχι. Και αυτό να συμπεριληφθεί στην αναθεώρηση του προγράμματος για το 2020. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Τζανίνη, κυρία Υπουργέ, πριν από την παρέμβασή σας στην αίθουσα αυτή μιλήσαμε για την ε, ανταγωνιστικότητα, για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος ε, είναι έτοιμος ε, να, να παράγει τα δικά μας περίπου τα προϊόντα, γιατί υπάρχουν πάντα πιο φτωχές χώρες από τις δικές μας. Άρα δηλαδή το μυστικό είναι να διατηρήσει κανείς στην Ευρώπη το know-how και ίσως όχι τόσο την παραγωγή. Ίσως αυτή να είναι η λύση. Άρα δηλαδή σωστό είναι αυτό που λέγεται για την ανάπτυξη, όμως αυτό που λείπει είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Δηλαδή οι επιχειρήσεις να έρθουν κοντά στα σχολεία. Κανονικά όταν μιλάμε για αυτό έχουμε πάντα κατά νου τους ε, ε, φοιτητές οι οποίοι κάνουν την εκπαίδευση στις επιχειρήσεις, αλλά να πάμε και αντίθετα. Οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για να εκπαιδεύουν εκείνους οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν επιχειρήσεις και όχι αντίστροφα όπως σας το είπα προηγουμένως. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μεταφέρουμε και το μεταποιητικό, τη μεταποιητική τεχνογνωσία, δηλαδή να επενδύσουμε έτσι ώστε να συμβεί και αυτή η προβολή της γνώσης αυτής. Κλείνω με μία ερώτηση το ευρωπαϊκό round table που τώρα πλέον έχει θεσμοθετηθεί εδώ στις Βρυξέλλες. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί κανείς να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της έρευνας ε, με βάση τις επιθέσεις που δέχεται η έρευνα αυτή από τις πολυεθνικές εταιρείες στην Ευρώπη. Κυρία Υπουργέ, αν έχει την καλοσύνη να μας απαντήσετε. και μία καταληκτική, ε, μία κατακλίδα πριν ολοκληρώσετε. Ξεκινώντας από το ερώτημα του κύριου Κάρεντς. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είναι γενική, αλλά στέκεται σε ένα σημαντικό θέμα. Πώς μπορεί να γίνει το Horizon 2020 ένα πραγματικό εργαλείο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικό όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τον ακαδημαϊκό χώρο, τα κρατη αλλά και για την κοινωνία. Δύο μεγάλες προκλήσεις. Πρώτον, να υπάρξει διεπιστημονικότητα. Το Horizon αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον της ε, κοινωνίας μας. Κλίμα, μετανάστευση που δεν είναι ένα εθνικό αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το να είναι κανείς διεπιστημονικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σημαίνει να προσπαθεί κάποιος να βελτιώνει τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα που εκ της φύσεώς τους είναι διεπιστημονικά. Αυτό είναι το πρώτο εργαλείο που βλέπω στην ε, ε, ημερήσια διάταξη και από την οπτική της Ιταλίδας Υπουργού. Και δεύτερον, να συνδυάσω ε, αυτά που ρωτήσατε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα το ιδιωτικό με το δημόσιο ώστε να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την ενέργεια που μπορούν να παράγουν. Στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά από ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα. Και αυτό πάει και σε κάτι που είπε ένας άλλος συναδελφός σας, δεν είμαι βέβαιη. Ο κύριο Ντεμπάκερ νομίζω, αλλά δεν είμαι βέβαιη. Ναι, εκεί. Μία από τις τρεις υποερωτήσεις που θέσατε πηγαίνουν, πηγαίνει και προς την κατεύθυνση που προσπάθησε ήδη να απαντήσω. Στον κύριο Κάρενς για το τεράστιο κενό το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της Ευρώπης αφενός και των άλλων μεγάλων εμπλεκομένων εκτός Ευρώπης σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα ότι ένα άλλο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, αλλά και για σας το Κοινοβούλιο, στην επόμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου, είναι η προσπάθεια να συνδυάσουμε τα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα με τα διεθνή, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς που διαθέτουμε για να προσελκύσουμε ταλέντα, ερευνητές εκτός από χώρες εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο που έχουμε για να και που πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με το τι κάναμε στο παρελθόν. Για τη δεύτερη ερώτηση του κ. Γκρίμπατσελ Συμφωνώ μαζί σας για το θέμα της εκπαίδευσης. Δεν μίλησα για την εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα συζητήσω με την αρμόδια επιτροπή σε δύο μέρες, οπότε δεν ήθελα να το θίξω σήμερα, αλλά εκμεταλλεύομαι την ερώτησή σας για να απαντήσω. Έρευνα, εκπαίδευση, ανάπτυξη είναι πολλές πλευρές του ίδιου νομίσματος. Our, ε, and our new... Πρέπει να προβάλλουμε τους στόχους μας και στον τομέα της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι η απάντηση στο δραματικό πρόβλημα που έχουμε, την ανεργία των νέων ιδίω. Να απαντήσω στα Ιταλικά μια και έχω τη δυνατότητα. Προς τον κύριο Ρόμπα. Αν η περικοπή του κοινοτικού προπολογισμού που έγινε στον τομέα της έρευνας είναι λάθος ή όχι. Ως έχουσα την Προεδρία της Ένωσης η απάντηση είναι μία ουδέτερη απάντηση που πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις που υιοθετήθηκαν και που είναι καρπός ε, διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, αν μου, θέτετε, αν θέτατε το ερώτημα αυτό υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργού Έρευνας, το θύμισε και ο Πρόεδρος ότι στο παρελθόν ήμουν πανεπιστημιακός, θα απαντούσα ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι σημαντική επένδυση πόρων στον τομέα της έρευνας. Οι συνάδελφοι τα Μπουράνο και Μπορέλη. Η εκπαίδευση ως στρατηγικός, στρατηγικό asset, στρατηγικό πλεονέκτημα. Προφανώς, ναι. Τα ιταλικά ζητήματα μπορούμε να τα συζητήσουμε αλλού, όχι εδώ. Πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καθοριστικό νομίζω οι δύο θέσεις του προπολογισμού που αυξήθηκαν και γι' αυτό υπήρξε και η μείωση που σχολιάσαμε προηγουμένως ήταν ακριβώς το Horizon 2020 για την έρευνα και τεχνολογία του Erasmus Sin που αφορά μία πολιτική κατάρτισης, την κινητικότητα των φοιτητών. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση του Κοινοβουλίου κατά βάση. Για τον κύριο Μπορέλη που μιλά για σχολείο και κατάρτιση, πρακτική κατάρτιση και ποιο εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αποφυγή μιας ηγεμονικής παρουσίας των μεγάλων ομάδων ομίλων που μπορούν να ασκήσουν προτεραιότητα, κατά προτεραιότητα ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι η πρόταση για ένα σωστό μοντέλο συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, όπως αυτό που, περιέβαλα, που περιέγραψα νωρίτερα για, την, για τις Joint Technology Initiatives, Δώδεκα δις νομίζω έχει βάλει η Επιτροπή Με ακούσατε, διακόπτει ο μιλήτρια. Μπορεί έλεγα να είναι ένα μοντέλο, αυτό το ΣΔΙΤ, ε, ιδιωτικό δημόσιο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τελευταία ερώτηση. του κύριου Τάλιτσκα που λέτε πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της καινοτομία πέραν του καταλόγου προτεραιοτήτων. Ξέρουμε ποιες προτεραιότητες εν γέννη. Έχουμε ήδη εφαρμόσει στον τομέα της έρευνας σωστά εργαλεία μέτρησης της καινοτομία και νομίζω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο Ίσως να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διεθνή επιτροπή που θα μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση βάσει ε, εγκεκριμένων benchmarks οροσίμων, αυτών δηλαδή μέσων που χρησιμοποιεί μια ομάδα ή μια επιχείρηση μεταξύ της, του ίδιου του έργου, δηλαδή του στόχου του έργου και του αποτελέσματος του έργου, που είναι ένας καλός τρόπος μέτρησης. Τι σημαίνει η καινοτομία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ah, yeah, yes, I already my, speech uh, how, uh, to what is a priority for Την ομιλία μου δεν ξέρω αν ανέφερα πόσο σημαντική είναι για την Ιταλική Προεδρία του να αναθεωρήσει βραχυπρόθεσμα την στρατηγική Ευρώπη 2020 με η έμφαση θα είναι στην προσπάθεια συνδυασμού των πραγματικού συνδυασμού μεταξύ των εθνικών και του ευρωπαϊκού προγράμματος. Όχι μόνο του, του Horizon 2020, αλλά και των διαφορετικών πόρων που δίνουν σαφείς καθηγητήρες γραμμές και παρέχουν τεράστια κονδύλια για την συνοχή, την κοινωνική καινοτομία και μια σειρά άλλων θεμάτων που προσπάθησα να αναφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που δώσατε και επίσης και σας ευχαριστούμε και για τη συζήτηση με την Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε κάθε καλό για τους επόμενους τέσσερις μήνες που δεν είναι και πολύ μακρά η περίοδος. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν και ως Επιτροπή Ήτρε αρμόδιοι για την έρευνα την καινοτομία και το διάστημα προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με την Ιταλική Προεδρία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη χρηματοδότηση όλων αυτών των πραγμάτων ε, που συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια τη Ιταλικής Προεδρίας. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε χρόνο για μας και σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κάθε καλό για το μέλλον. Ε, well, thank you. Dear friends, dear Αγαπητοί φίλοι, ας πάμε λοιπόν τώρα στο πραγματικά τελευταίο θέμα της συναντησής μας που είναι διάφορα. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα σε αυτό το θέμα. Επόμενη λοιπόν συνάντηση, πολύ σημαντικό, 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες και 25 Σεπτεμβρίου 9 με 12.30 και τρεις ε, με 6,5. Δηλαδή ε, θα κρατήσει περισσότερο η συνεδρίαση εκείνη από τη σημερινή. Κάθε φορά λοιπόν ε, θα συναντιόμαστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα έχουμε όλο και πιο πολύ δουλειά να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.